Allora, ε, Ξεκινήσουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Να ενημερώσω την Επιτροπή για τις ε, συστάσεις των ε, συντονιστών από την χθεσινοβραδινή συνεδρίαση, οι οποίες ελπίζω, οι οποίες ελπίζω πως θα εγκριθούν. Πρώτα απ' όλα, αναθεώρηση του άρθρου 116 του κανονισμού του Συμβουλίου θα αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης από το ΕΛΚ. Αυτό για την ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου κατόπιν για τις εμπορικές ε, συμφωνίες τρίτον αίτημα για ερμηνεία του, άρθρου 50 του κανονισμού για συνδεδεμένες επιτροπές και για το πώς δύο επιτροπές μπορούν να υποβάλουν απευθείας. Σας σταλεί επιστολή από τον Πρόεδρο. Τέταρτο. για την εξέταση της διοργανικής συμφωνίας με το Συμβούλιο για κάποιες πτυχές της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας, η ομάδα των Πρασίνων θα, έχει, θα καθορίσει τον εισηγητή και θα ζητήσουμε ο εισηγητής να συμμετέχει στην ομάδα των διαπραγματευτών. Πέμπτον, από τις 24 έως τις 26 Μαΐου μία αποστολή έξι μελών από την Επιτροπή Συνταγματικών Επιθέσεων, δύο από το ΕΛΚ, δύο σοσιαλιστές, μία, ένας από την ΚΟΕΚ θα επισκεφθούν την Πολωνία. Θα το οργανώσουμε με τον κύριο Ταρκόφσκι, ο οποίος θα μας δώσει ίσως σήμερα κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες ε, στη διάρκεια της συνεδρίας της επί του θέματος. Έκτον, θα ζητήσουμε να ε, εκπονηθεί μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουν κάποια θέματα μονομερώς ε, τα κράτη-μέλη με το Συμβούλιο και ο κύριος Σταρκόφσκι είναι αυτός ο οποίος θα δει τι θα γίνει και πώς θα πρέπει να ερμηνεύσουμε τον κανονισμό. Θα πρέπει να δούμε το, ε, τι γίνεται με αυτή την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή ΑΦΚΟ θα ζητήσει από τον κύριο Σάγερ να ε, δει τι θα γίνει με τη διαδικασία ε, συνταγματικής μεταρρύθμισης στην Ουγγαρία. Θα εξετάσουμε και τη μελέτη που έχει ξεκινήσει για την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και για τις αναφορές. Αυτά επί τη βάση συστάσεων που θα δώσει ο κύριος Χέφρεν στην Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και για να δούμε τι θα γίνει. Δέκατον, θα ενημερώσουμε την Επιτροπή Αναφερών ότι δεν μπορούμε να δώσουμε καμία συνέγεια στην ε, αναφορά 08010 διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα για να υιοθετηθούν τα μέτρα τα οποία ζητούνται. Η Επιτροπή θα ζητήσει από τον ε, θεματικό τμήμα για τις μελέτες για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πολιτικό κόμμα σε ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδικασίες, ε, υποψηφιότητες ε, και ούτω καθεξής, εκλογικά δικαιώματα και συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πρόεδροι σε τρίτες χώρες και πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε χώρες της Ένωσης. Μία τέταρτη μελέτη σε γραπτή πρόταση η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 20 Μαρτίου και τέλος ο συνάδελφος Μέντες Δεβίγκο ζήτησε και οι, συγητές, ε, οι το δέχτηκαν και εγώ σας προτείνω μια έκτακτη συνεδρίαση για τις 22 Μαρτίου το απόγευμα στο, στις Βρυξέλλες για να εξετάσουμε για άλλη μια φορά ως Επιτροπή το θέμα της μεταρρύθμισης της συνθήκης, ε, το άρθρο 136, αυτό το διαβόητο ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει τόσο καιρό. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις του Προέδρου, δεν ξέρω αν υπάρχουν παρατηρήσεις, αλλιώς ε, θεωρούμε ότι εγκρίνονται από την Επιτροπή μας, ο κύριος Μέντε Δεβίγο. Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση που μόλις κάνατε έγινε για να μπορέσουμε να ακούσουμε τους κυρίους ε, Μπρόκ και Γκουαλτιέρη πριν από την Ολομέλεια ε, και την ψηφοφορία για να μπορέσουν να μας πούν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που έκαναν με την εντολή που τους δώσαμε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων την προηγούμενη εβδομάδα πριν από την Ολομέλεια, λογικά θα πρέπει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να ακούσει ε, από τους συζητητές ε, τι ε, αποφασίστηκε για να το γνωρίζουν και όλες οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Γνωρίζετε ότι στις Ολομέλειες της Βρυξέλλες είναι πολύ σύντομες χρονικά η συνεδρίαση των πολιτικών ομάδων. Επομένω, καλό θα ήταν να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε και αν μπορούμε ε, εμεί στην Επιτροπή να διαβιβάσουμε στι πολιτικέ ομάδε ε, τι ακριβώ συμβαίνει. Αυτή είναι η πρόταση και σα ευχαριστώ που την εγκρίνατε. Ο κύριος Γκολτιέρη. Ε, εγώ δεν είμαι κατά της πρότασης του κυρίου Μέντες ο πρόεδρος ε, θα αποφασίσει. Οι συντονιστές ε, ήταν υπέρ. Τώρα ε, εμείς θα πρέπει να το διαβιβάσουμε στην Επιτροπή και μπορούν κάλλιστα κάποιος να έχει ένσταση. Δεν βλέπω καμία ένσταση βέβαια. Θα συνεδριάσουμε λοιπόν το απόγευμα της 22ης Μαρτίου για να δούμε τι αποφασίστηκε διαστόματος στον κύριο Μπλέκ και Γκουαλτιέρη. Να περάσουμε τώρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης για σήμερα το πρωί. Καταρχάς έχουμε την έκθεση του συναδέλφου Νταφ για την ε, τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ κύριε Νταφ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Και σας ευχαριστώ για την επιμέλεια που δείξατε. Ε, με το να καταθέσετε αρκετές ε, τροπολογίες στο ψήφισμα για τις προτινόμενες αλλαγές ε, στη συνθήκη. Όπως ξέρουμε είναι πολύπλοκη η δομή και άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να υπάρχει μια συνοχή και στα τρία αυτά μέσα του προτινόμενου ψηφίσματος, της συνθήκης και του νομοθετήματος. Θα ήθελα να αναφέρω τέσσερις τροπολογίες ε, που κατέθεσα εγώ. Η πρώτη είναι η παριθμόν 25 η οποία έφιστα την προσοχή μας στο γεγονός ε, πως έχουμε επίσημη νομοθετική πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και άρα ε, εμπίπτει στο πρωτόκολλο περί εθνικών κοινοβουλίων και θα πρέπει να το παραπέμψουμε μετά τη συμφωνία στην Ολομέλεια στα εθνικά κοινοβούλια για τον έλεγχο της ε, επικουρικότητας. Κατόπιν, στην τροπολογία 81, ζητάω από την Κομισιόν να καταθέσει νωρίτερα την ε, πρόταση κανονισμού για να ενισχύσει τη Eurostat. σε σχέση με την ε, συνοχή και την συγκρισιμότητα των των ε, εθνικών στοιχείων. Κατόπιν στην 112 προτείνω ε, για, την, ε, για τον τύπο Σαβαρίν Λεμεσούρ για την φθήνουσα αναλογικότητα θεωρώ πως θα πρέπει να δούμε το εάν θα συμφωνηθεί τελικά ή όχι ε, μαθηματικός τύπος καθώς οπωσδήποτε βεβαίως ε, θα διευκολύνει ε, την υπερασπιστική γραμμή μας στα δικαστήρια εάν μας κατηγορήσει κανείς πως παραβιάζουμε την φθήνουσα αναλογικότητα εάν αλλάξουμε τον αρχικό τύπο ο οποίος ακόμα δεν έχει ε, γίνει νόμος σύμφωνα με αυτό το οποίο πρότεινα. Για το 136 ε, εδώ πέρα προτείνω τον λεγόμενο συμβιβαστικό τύπο του Cambridge. Ε, θα τα δούμε όλα αυτά ξανά στο τέλος. Κάποια σχόλια τώρα για τις α, ε, τροπολογίες κλειδιά, συνάδελφοι. Βεβαίως πάντα υπό την επιφύλαξη των πενιχρών γνώσεών μου στα γερμανικά. Ε, δεν θα έχουμε νομίζω τις μεταφράσεις ε, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ατυχές αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει όσο πιο συνοπτικά μπορώ επί των τροπολογιών αυτών ε, και όπως τις έχω καταλάβει να πω τα εξής. Ο κύριος Σέφλιν επανέρχεται στην οδηγία 93-109 και σωστά τονίζει την σημασία ε, αναθεώρησης της. Θα του έλεγα απλά πως το Κοινοβούλιο έχει ήδη τοποθετηθεί. Μπορούμε να μεταβάλουμε άποψη, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς ε, ως προς το τι ακριβώς κάνουμε. Υποψιάζομαι πως ο Επίτροπος Σεφτσεβιτς θα τοποθετηθεί από αυτό. Ε, ζητάμε μια αναδιατύπωση τρόπον Α της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Σέφλιν γενναία προτείνει να συνταχθεί, να συνταχθούν εκλογική ε, κατάλογη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι να πω, καλή τύχη εύχομαι. Ε, κύριος Κουαλτιέρη προτείνει να αλλάξουμε τη συνθήκη και να πούμε πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει με συνένεση και στις προτινόμενες αλλαγές και όχι με ομοφωνία όπως τώρα. Καλή τύχη και σε αυτόν εύχομαι. Ε, θα πω πως εάν κάνουμε κάτι τέτοιο α, οπωσδήποτε θα χρειαστεί δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, και τότε καλή τύχη στους Βρετανούς. Um, uh, uh, um uh, Οι Τροπολογίε τώρα 70 και 71 ΕΛΚ και Σοσιαλιστών έχουν ως στόχο να μετατρέψουν αυτό το οποίο προτείνω εγώ δηλαδή μια διεθνή λίστα εκλογικών συστημάτων από πρώτη μισιακή σε κλειστή δηλαδή αντί να μπορεί να επιλέξει υποψήφιο σε μια λίστα ο ψηφοφόρος η μόνη επιλογή θα είναι να επιλέξει ένα μπλοκ το οποίο θα έχει προκαθοριστεί από το πολιτικό κόμμα είμαι κατά και πρέπει να είμαι ειλικρινής θεωρώ πως θα μειωθεί έτσι η ισχύ της μεταρρύθμισης δεν θα μπορέσει να ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια ο πολίτης την οποία χρειαζόμαστε για να ενθαρρύνουμε την συμμετοχή στις εκλογές σε δίθνες Η επιλογή μεταξύ προσωπικότητων και εθνικότητων θα αποτελέσει παράγοντα ενθάρρυνσης ε, της συμμετοχής ψηφοφόρων ε, στην ε, δεύτερη ψηφοφορία για την ε, διεθνή λίστα. Αν δεχτούμε την πρόταση σοσιαλιστών και ΕΛΚ είναι αντικίνητρο για την προσέλευση και θα δώσουμε και πάρα πολύ μεγάλη ισχύ στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Εντάξει, να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη αυτών των κομμάτων εγώ είμαι υπέρ ξέρετε, αλλά το να τους δώσουμε την εξουσία να προκαθορίσουν έναν κλειστό κατάλογο υποψηφίων μου φαίνεται ένα λυπηρό βήμα προς τα πίσω. Η πράσινη, ο Γκέλτ Χέφνερ, ο οποίος απουσιάζει περίεργος, προτείνει νομίζω να πάρουμε 25 ευρωβουλευτές από τους 751 ε, που είναι τώρα ε, κάτι το οποίο νομίζω είναι πολιτικά αδυνατόν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ξαφρίσουμε 25 βουλευτές από το τωρινό μέγεθος του σώματος δεν γίνεται αυτό η κυρία Μπελιέ θέλει να αυξηθούν οι 25 στους 27. Αντιλαμβάνομαι γιατί θέλει, αλλά νομίζω πως θα δημιουργήσει σύγχυση, θα δημιουργήσει την εντύπωση πως κάθε κράτος μέλος μπορεί να έχει έναν παραπάνω ευρωβουλευτή από αυτό το πείραμα. Και δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βρετανός συνάδελφος από το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα θέλει περιφερειακές εκλογικές ε, περιφέρειες στα κράτη-μέλη και εδώ ακολουθούν, τον ακολουθούν και κάποιοι Φιλανδοί και Σκανδιναβοί συνάδελφοι που θα ήθελαν οι αυτόνομες περιοχές όπως η νήσι Φιόλεντ να εκπροσωπούνται απευθείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο σε μια ενιαία εκλογική διαδικασία. Και είναι αρμοδιότητα της Φιλανδίας, παραδείγματος χάρη, να οργανώσει τα εσωτερικά της όσον αφορά τις αυτόνομες ε, περιοχές. Η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών, η οποία επίσης απουσιάζει, περιέργως, θέλει τη διαγραφή των ε, διεθνών λιστών όπως ξέρουμε οι κύριοι Γκουερέρο και Γκουαλχέρη προτείνουν ε, και δομικές και ουσιαστικές αλλαγές στις αλλαγές που προτείνω στο πρωτόκολλο <coughs> περί ασυλίων, και προνομίων αυτό πρέπει να γίνει στο πρωτογενές δίκαιο δηλαδή η ιδέα το ότι με έναν κανονισμό θα ξεκαθαρίσουμε τις λεπτομέρειες δευτερογενής νομοθεσία δηλαδή νομίζω δεν επαρκεί για να διασφαλίσουμε τις ασυλίες ενός ευρωβουλευτή στο υπερεθνικό επίπεδο. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Ο κύριος Γκουαλτιέρη και πολλοί Ιταλοί συνάδελφοι προτείνουν πως ε, όσοι έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα δεν θα πρέπει να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εθνικές προσεγγίσεις ε, διαφέρουν εδώ πέρα, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Ε, μπορεί να αποδεκατήσει βεβαίω και το σώμα, δεν ξέρω. Ε, εν πάση περιπτώσει να το συζητήσουμε. Όσον αφορά το μαθηματικό τύπο θα ήθελα να μείνουμε στην απόφαση που είχαμε λάβει επί της αρχής για να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε σε ένα μαθηματικό τύπο που θα είναι διάφανος, αποτελεσματικός, συνταγματικός και νομικά και να στέκει νομικά στα δικαστήρια. Γιατί βεβαίω όσοι θέλουν να σταματήσουν αυτή την προσπάθεια Α σκεφτούμε τι, τι θα κάνουν. Και εμείς πρέπει να σκεφτούμε βεβαίω τι θα κάνουμε για να υπερασπίσουμε το κοινοβούλιο κατά της κατηγορίας ε, που προέρχεται παραδείγματο χάρη και από το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, πως, είμαστε, πως παραβιάζουμε την συνθήκη. Θεωρώ λοιπόν πως ο συμβιβασμός του Κέμπριτζ που ζητήσαμε, ο μαθηματικός τύπος αυτός και αποτελεί αντικείμενο συνένεσης μεταξύ διαφορετικών μαθηματικών που ανταγωνίζονταν στο παρελθόν νομίζω πως εκπληρώνει και τους περιορισμούς της συνθήκης περί κατοφλίου, οροφής και μεγέθους και σέβεται την αρχή της ευθύνουσας αναλογικότητας. Και άρα εκπληρώνει τους ε, φιλόδοξους ε, στόχους μας. Ε, ένα σύστημα λοιπόν το οποίο συμφωνούμε πως θα πρέπει να είναι εύρωστο, να διαρκέσει για πολλές θητείες του Κοινοβουλίου και να είναι ανεξάρτητο από την πολιτική. Και θέλω να το τονίσω αυτό το τελευταίο. Μπορούμε βεβαίως να επιστρέψουμε στο πολιτικό παζάρι που είχαμε στο παρελθόν. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε για την αμεροληψία αυτού του παζαριού. Την αμεροληψία ως προς τις πολιτικές προτιμήσεις. πρόταση του Τζέρελτ είναι ένας παραβολικός τύπος που επιλέγει αυθαίρετα κάτι και χρειάζονται βεβαίως αυτά τα τρία τεστ που είπαμε για να ε, επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και θα είναι λιγότερο αναλογικός τελικά από τον συμβασμό του Κέμπριτζ. Η τελική έκθεση συμπτωματικά ε, του Cambridge ε, σας έχει ήδη διανεμηθεί και νομίζω αξίζει να την διαβάσετε με προσοχή. Ως για το τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ να ακούσω τους συναδέλφους. Εγώ προτείνω την επόμενη Τρίτη το απόγευμα γύρω στις 5 να συναντηθούμε οι σκιώδει ε, εισηγητές και θα καταθέσω μια συμβιβαστική πρόταση βασισμένη στη συμβαστική λύση του Κέμπριτζ με σταδιακή εισαγωγή ε, σε, διάφο... σε πολλές θητείες και θα σας εξηγήσω πώς θα γίνει αυτό. Ζητώ επίσης μια ειδική συνεδρία της Επιτροπής μας στο Στρασβούργο το πρωί της 7 για να δούμε τι θα έχει συμβεί και στις ομάδες μας ε, στο Στρασβούργο και βεβαίω ε, το πρόγραμμα είναι ακόμα να ψηφίσουμε στις 19 του επόμενου μήνα όπως είχαμε συμφωνήσει. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Νταφ. Έχω πολλούς εγγεγραμμένους, ε, αλλά στις 10 θα πρέπει να ψηφίσουμε για την έκθεση Γιαννάκου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να περιοριστείτε σε τρία λεπτά το πολύ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Ντάφ για τη συναρπαστική και εξαιρετικά σημαντική έκθεση. Με πολλά από αυτά δεν έχουμε πρόβλημα. Οι υπερεθνικές λίστες και τα λοιπά η μόνη μου επιφύλαξη είναι πως αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα περί ήμι ανοιχτών ληστών και να μην δώσουμε πάρα πολύ εξουσία στα κόμματα, αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι πως στην περίπτωση αυτή η δυνατότητα να παρισφρήσει η εθνική εκλογική συμπεριφορά υπάρχει. Οπότε εγώ είμαι υπέρ ε, Τη κλειστή λίστα, παρά το ότι είναι λιγότερο δημοκρατική όσον αφορά το εάν η, η μη ανοιχτή λίστα θα κινητοποιήσει λιγότερο τους ψηφοφόρου, εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος. Τα εθνικά στοιχεία πάνε και προς τι δύο κατευθύνσεις. Καμιά φορά ναι, καμιά φορά όχι. Οπότε εγώ λέω πω θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις κλειστέ λίστε παρά τα αντίθετα επιχειρήματα. Ο εκλογικό κατάλογο τον οποίο ανέφερε ο κύριο Ντάφ Εάν είναι να έχουμε υπερεθνικές λίστες, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και το να έχουμε εν πανευρωπαϊκούς ευρωπαϊκούς ε, καταλόγους. Βεβαίως δεν είναι πολύ ικανοποιητικό το σύστημα. Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που υπάρχουν, ε, είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια. Από την άλλη, δεν θα έλεγα πως είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά οπωσδήποτε βοηθάει πάρα πολύ για να λειτουργήσουν ε, επιτυχώς οι υπερεθνικές λίστες. Το πραγματικό πρόβλημα το οποίο έχουμε εμείς βεβαίως αφορά το μαθηματικό τύπο. Εάν δείτε την έκθεση που τουλάχιστον εγώ βρήκα στο γραφείο μου σήμερα το πρωί, οι χώρες μέσου μεγέθους αδικούνται. Ο συμβασμός του Cambridge μπορεί να είναι αποτελεσματικός και να στέκει στα δικαστήρια και μαθηματικά να είναι βεβαίως θαυμάσιος, αλλά οι πολιτικές του συνέπειες για τις μεσαίες χώρες είναι απαράδεκτες, καθώς πλην της Γερμανίας εποφελούνται οι μεγάλες χώρες. Δεν νομίζω λοιπόν πως είναι τέλεια λογική για να ξεκινήσει μια φιλοευρωπαϊκή εκστρατεία. Μάλλον το αντίθετο. Θα ξεκινήσει μια αντιευρωπαϊκή εκστρατεία. Δεν ξέρω εάν οι Ούγγροι ε, ψηφοφόροι μου θα βγουν ε, και θα τραγουδούν στους δρόμους αν μάθουν πως πάνε από τις 20 έδρες στις 17. Ε, είναι απαράδεκτο. Αντιλαμβάνουμε βέβαια στην πολιτική σημασία και χρησιμότητα το να έχουμε έναν τύπο ο οποίος θα στέκει στα δικαστήρια και πράγματι έτσι τελειώνει το πολιτικό παζάρι το οποίο έχουμε συζητήσει αλλά νομίζω πως οι πολιτικές συνέπειες είναι τέτοιες ε, που δυστυχώς δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε και κάποια πραγματάκια ακόμα συνολικά, δηλαδή κάτι αναφορές για εθνικές μειονότητες και τέτοια, δεν ξέρω, νομίζω πως θα πρέπει να μιλήσουμε για όλες τις μειονότητες. Και πέρα από αυτό η έκθεση είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ τον κύριο Ντάφη και θα σταματήσω εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που πρέπει να σας περιορίσω, αλλά πρέπει να το κάνω. Ο κύριος Γκολτιέρη τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο αριθμός των τροπολογιών ε, στην έκθεση επιβεβαιώνει πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα αυτό και το γεγονός ότι ο κύριος Νταφ δεν μας έχει προτείνει μια κοινότυπη έκθεση, αλλά μια έκθεση η οποία δημιουργεί και το έναυσμα για να σκεφτούμε και να δώσουμε και μια ανάσα. Εγώ θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τις τροπολογίες της ομάδας μου, ομαδοποιώντας τις ανά σημείο. Καταρχάς το θέμα του υπερεθνικού καταλόγου. Ένα θέμα το οποίο είναι διαφιλονικούμενο. Δεν σας το κρύβω άλλωστε. και υπάρχουν αρκετές ενδείξεις υπέρ, αλλά ταυτόχρονα και πολυάριθμα προβλήματα. Η απόφασή μας βέβαια ήταν να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση, η οποία είναι βασική πρόταση της έκθεσης DAF. Ωστόσο, θέλουμε να προτείνουμε μια τροπολογία ώστε να μην υπάρχει καμία αναφορά στις προτιμήσεις, ακόμα και αν πρόκειται για την ε, μια ανοιχτή μέθοδο, για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε διαφορετικές πραγματικότητες σε εθνικό επίπεδο και να υπάρχει και ε, ο κατάλογος προτίμησης, ο οποίος ε, θα είναι και κατάλογος ανάλογα με το μέγεθος ε, των ε, κρατών στον οποίο συμμετέχουν υποψήφοι, στο, του οποίου η πίκο είναι υποψήφοι. Ε, εμείς αποφασίσαμε να μην υπάρχουν προτιμήσεις, αυτό προτείνουμε. Όσον αφορά τώρα το μαθηματικό τύπο, Σαφώ η πρόταση ανταποκρίνεται στα τρία κριτήρια που μα υπέδειξε ο κύριο Σταφ και εγώ προσωπικώς τη βρίσκω λογική και θεωρώ ότι ανταποκρίνεται και σε ένα αφηρημένο κριτήριο ε, μεγαλύτερης αναλογικότητας ακριβώς διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο του άμεσου εκπροσώπου των πολιτών και η εκπροσώπηση των κρατών μελών μετατοπίζεται περισσότερο προς το Συμβούλιο και επομένως όπως είχαμε προβλέψει η διάρκεια του μαθηματικού τύπου και το γεγονός ότι επιλέγουμε μεταξύ των διαφόρων συστημάτων προκειμένου να είναι πιο αναλογικό το σύστημα. Καταρχάς υπάρχει το Fix Pro που είναι το πιο αναλογικό με βάση 5 όμως αυτή την περίπτωση, δηλαδή ακόμα και πιο, ο πιο ακραίος συντελεστής επιλέγεται εδώ. Θέλουμε να έχουμε δηλαδή τέτοια αναδιανομή που από πολιτικός και τεχνικό κης ε, άποψης να είναι δύσκολο να βρούμε πλειοψηφία που θα υποστηρίξει αυτή την πρόταση. Εμείς θέλουμε να προτείνουμε ένα λακτικό δρόμο, φιλόδοξο, που ε, ζητά και αλλαγή τη συνθήκη. Ο κύριο Ντάφ μου ευχήθηκε να το πετύχω, αλλά εγώ σας διευκρινίζω ότι ούτως ή άλλως προτείνουμε μεταρρύθμιση τη συνθήκη με τον κατάλογο αυτό που θα οδηγήσει σε πολλές αιτήσει για ε, δημοψηφίσματα. Αφού λοιπόν ούτως ή άλλως ακολουθούμε την άγουσα της μεταρρύθμισης της συνθήκης και θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσει ε, να το τμήμα της συνθήκης που απευθύνεται στην ε, κατανομή του Κοινοβουλίου να προσπαθήσει να το κάνει πιο συνεκτικό ω προς τη συνθήκη. Η συνθήκη της ε, Λισαβόνα αλλάζει και λέει αντί για εκπρόσωπο, ότι το Κοινοβούλιο αντί για εκπρόσωπο των κρατών μελών είναι εκπρόσωπο των πολιτών και το Συμβούλιο είναι ο εκπρόσωπος των κρατών μελών. Επομένω, εδώ υπάρχει αντίφαση μεταξύ των αρχών της συνθήκης και της ίδιας της συνθήκης. Εάν λοιπόν ούτω ή άλλω προσπαθούμε να αλλάξουμε τη συνθήκη, όπω προτείνει ο κ. Νταφ και φαίνεται ότι συμφωνούν και οι περισσότερε πολιτικέ ομάδε αυτή τη στιγμή δέχονται την αρχή αυτή του υπερεθνικού καταλόγου, ε, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να πάμε στην πηγή όλων των προβλημάτων. Και το γεγονός είναι ότι η σύνθεση του Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να επαφίεται μόνο στο Συμβούλιο, αλλά θα πρέπει να συναποφασίζεται μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η έννοια τη τροπολογία μου δεν είναι μια τροπολογία η οποία απλώς λέει όχι στο μαθηματικό τύπο, αλλά ε, προκαλεί και σε μια νέα μάχη που ίσως θα μπορέσει να βρει και το Κοινοβούλιο ενωμένο σε αυτό το ε, ζήτημα, παραταγμένο κατά του Συμβουλίου. Υπάρχουν και κάποιες τροτοβουλίες, ο κύριος Χέφνερ προτείνει αυτό τον παραβολικό τύπο, ο οποίος είναι πιο βιώσιμος από το fix prop, αλλά εμείς αποφασίσαμε να μετατοπίσουμε το βάρος στη διαδικασία και όχι τόσο στη φύση της ε, ανακατανομής των εδρών. Υπάρχει τώρα μια ακόμα σειρά τροπολογιών η οποία συσχετίζεται με αυτό που μόλις σας είπα, ε, τη δική μου τροπολογία. Κύριε Γουαλτιέρη, διακόπτει ο Πρόεδρος, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, θα είμαι λακωνικός. Προσπαθούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε την ίδια λογική που ακολουθούμε και με το θέμα της ε, σύνθεσης και για άλλες πτυχές για τις οποίες και πάλι υπάρχει μία νομοθεσία η οποία έχει μείνει στη λογική που είχαμε πρώτης συνθήκης Λισαβόνας. Ε, αντί να επιλέξουμε τώρα την ημερομηνία των επόμενων εκλογών, θα πρέπει να πούμε ότι την ημερομηνία των επόμενων εκλογών θα πρέπει να την αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μην σταθούμε στις ε, λεπτομέρειες για τους ε, νόμους και τις δυνατότητες και το περιθώριο ευελιξίας. Απλώς θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτό θα πρέπει να το συναποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτές τις αποφάσεις στο Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο είναι ο άμεσος εκπρόσωπος των πολιτών. Τέλος, δύο σύντομε παρατηρήσεις και ζητώ συγγνώμη, θα είμαι λακωνικός. Το πρώτο είναι ότι διαπίστωσε ότι αρκετοί συνάδελφοι, όχι αυτοί μόνο που ανέφερε ο κύριο Νταφ, αλλά και κάποιοι άλλοι εμέσω αναφέρονται σε διάφορα άρθρα και όχι στο άρθρο 2 και τα περιφερειακά ε, συμβούλια, περιφερειακό σώμα. Μου φαίνεται ότι οι παραπομπέ αυτέ ε, είναι αδόκιμε, διότι υπάρχει το άρθρο 1 σημείο 2 ή μάλλον, στο άρθρο 1.1 λέγεται σαφώς ότι μπορούμε να καθορίσουμε. Έκανα λάθο παράθεση, λέει ο, ο αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να δημιουργήσουμε περιφερειακά συμβούλια χωρίς να αγγίξουμε τον αναλογικό χαρακτήρα της ψήφου. Και αν δεν ε, πειράξει κανεί αυτή την αρχή και κανένα δεν προτείνει να την αλλάξουμε, δεν υπάρχει νόημα να πάμε σε άλλα σημεία τη νομοθεσία και, να και να εισαγάγουμε στοιχεία για τα περιφερειακά ε, συμβούλια που θα μπορούσαν να έρθουν σε αντίθεση με την αναλογική αρχή της ψηφοφορίας. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή διαφορετική κατανομή στην οργάνωση της λίστας, ε, μπορεί να είναι τοπικές, ε, περιφερειακές, αναεκλογική περιφέρεια. Ε, αλλά δεν θα ε, υπερβαίνουν την ε, εθνική αναλογικότητα της κατανομής των εδρών, γιατί αυτή είναι μια αρχή η οποία είναι υπέρ όλων των υπολείπων και κανένας δεν θέλει να την αλλάξει και κανένας δεν θέλησε και να την αλλάξει. Και τέλος, ε, μια τροπολογία για τους καταδικασμένους. Υπάρχουν τρεις ομάδες αδικημάτων, οι οποίες έχουν σχέση και με τη δημόσια τάξη, εργανομένο έγκλημα, διαφθορά και υπάρχουν και υψηλέ ποινέ και υπάρχουν και μια κατηγορία ποινών ε, όπου υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ε, Εμεί επιλέξαμε ως κριτήριο δηλαδή αδίκημα για το οποίο ε, η ποινή είναι άνω των τριών ετών. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για αυτούς του οποίους δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ πλήρως πως αυτή η έκθεση του συναδέλφου του Άντριου Ντάφ είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά υπάρχουν κάποιες επιλογές που είναι απολύτως απαράδεκτες. Πρώτα απ' όλα να πω πως αντιλαμβάνομαι την επιλογή της αναλογικότητας, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι το ότι ο Άντριου Νταφ θεωρεί πως 27 κρατη στην υπερεθνική λίστα είναι κίνδυνος γιατί υπάρχει ο κίνδυνος εθνικής ε, προσέγγισης. Μα με την προτιμησιακή ψήφο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εθνικής προσέγγισης στην ψηφοφορία. Είναι αντιφατικό να απορρίπτουμε τους 27 και μετά να επιλέγουμε ε, το σύστημα. Κατόπιν, να σας πω τι, κατά τη γνώμη μου, εκπλήσει το ότι έχουμε εδώ αυτή τη φόρμουλα για την οποία για πρώτη φορά απορρίπτω το ότι πρόκειται περί συμβιβασμού. Όχι, δεν πρόκειται περί συμβιβασμού μεταξύ ουδήποτε. Εδώ κάποιος αυθαίρετα επέλεξε αυτή τη φόρμουλα. Όχι, όχι, εμείς Πορτογάλοι δεν ε, θέλουμε κανέναν συμβασμό. υπάρχει όταν υπάρχει συμφωνία για κάτι. Και αυτό το οποίο ανέφερα είναι το ότι θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει τέτοιου υπηρεσία και κατόπιν να προσπαθούμε να πετύχουμε κάποια λύση. Αλλά όχι, δεν πρόκειται περί συμβασμού για οτιδήποτε. Επομένω, 100% απορρίπτω ακόμα και τη διατύπωση. Και επίση, απορρίπτουμε το ότι έχουμε αυτή την ουδέτερη διατύπωση, ουδέτερη φόρμουλα. Δεν υπάρχουν φόρμουλες ουδέτερες. Διαφορετικά συστήματα υπάρχουν. Και είναι σαφές ότι θέλετε να δώσετε στις μεγάλες χώρες, μεγαλύτερο ειδικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλετε να εξουθενώσετε τις μεσαίες χώρες. Πορτογαλία, Σουηδία, Τσεχία κλπ. Πρόκειται για μια κατάσταση απαράδεκτη σε αυτή την περίπτωση. Επομένως δεν πρόκειται περί ουδέτερης επιλογής. Δεν υπάρχουν δεύτερες επιλογές. Και εκεί που αναφέρατε το... The... Αναφέρετε το συνταγματικό δικαστήριο. Έχω να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση και συγκρισιμότητα μεταξύ της ευρωπαϊκής πολιτικής ισορροπίας δυνάμεων και της γερμανικής. Αλλά όμως ακόμα και για τη Γερμανία και δεν λέω για την Βουλή αλλά για τη Γερουσία ακόμα και εκεί υπάρχουν διαφορετικά συστήματα ψηφοφορίας που δεν είναι αναλογικά. Και το ίδιο και με το Συμβούλιο, σε αντίθεση με το Κοινοβούλιο. Υπάρχει διαφορετικό σύστημα. Άρα, το προτινόμενο είναι απαράδεκτο. Άντριο Ντάφ, έχω να πω ότι η συζήτηση είναι πάρα πολύ εμβριθής, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά όπως μας ευχαριστήκες και εσύ καλή τύχη, σου εύχομαι και εγώ καλή τύχη με αυτό το μαθηματικό τύπο, αυτή τη φόρμουλα. Χέφνερ, παρακαλώ και εσείς σύντομος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ βλέπω πως πραγματικά εδώ πέρα ο Άντριου Νταφ ε, έχει προσεγγίσει το θέμα πολύ αποφασιστικά και εδώ πέρα υπάρχουν δύο μεγάλοι στόχοι. Το ένα είναι να γίνουν ευρωεκλογέ πιο ευρωπαϊκές και να γίνουν και πιο δημοκρατικές. Υποστηρίζω την ιδέα μιας ε, ευρωπαϊκής εκλογικής περιφέρειας για 25 βουλευτές και να δώσουμε έτσι την δυνατότητα στους πολίτες να μην ψηφίζουν μόνο συμπατριώτες τους, ανθρώπους από το δικό τους κράτος μέλος, αλλά και βουλευτές από μια πανευρωπαϊκή λίστα. Υποστηρίζω επίσης την ιδέα η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει μέσω, μιας, ε, μέσω ενός ενιαίου τύπου και να μην μπορεί πλέον να υπάρχει υποψία αυθαιρεσίας, ε, παζαριών κτλ. Ε, νομίζω πως αυτό θα μας βοηθήσει ε, στην συνταγματική και πολιτική συζήτηση και στα κράτη-μέλη και στα δικαστήρια. Θέλω να πω επίσης κάτι άλλο. συγγνώμη για το, το λαιμό μου πρέπει ε, να εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά πρώτα το νομικό και συνταγματικό ζήτημα για να είναι τελείως άμεμπτο και δεύτερον πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ε, μια λύση η οποία θα δημιουργήσει λιγότερες αντιστάσεις και θα έχουμε τους περισσότερους συμμάχους. Δηλαδή θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες υιοθέτηση με την κατανομή εάν μείνουμε κοντά στην τωρινή κατάσταση και λιγότερες δυνατότητες να απομακρυνθούμε πάρα πολύ. Θα θυμάστε πως ρώτησα τρεις φορές στην ακρόαση ε, τα της κατανομής των εδρών γιατί βλέπω σοβαρά προβλήματα και ρώτησα εάν γίνεται κάτι διαφορετικό και τρεις φορές μου είπαν πως δεν γίνεται διαφορετικά. Καθίσαμε δύο μέρες ε, Προσπαθήσαμε με διάφορους ε, τύπους, ε, δεν καταλήγαμε σε καμία άλλη μαθηματική λύση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπέβαλα διαφορετικό τύπο. Όχι γιατί θέλω να αναγκάσω την Επιτροπή να υιοθετήσει τον δικό μου τύπο, αλλά γιατί πάντα ε, αυτό το οποίο βρίσκω εκνευριστικό στην πολιτική είναι να λέμε αυτός είναι ο δρόμος, ο μοναδικός και δεν υπάρχει άλλη λύση. Όχι, υπάρχουν και άλλοι ε, τρόποι και έχω παρουσιάσει εδώ πέρα σε μια καμπύλη, μια κατανομή και βλέπετε πως ειδικά οι μεσαίες χώρες χάνουν ε, πολύ λιγότερες έδρες ε, με αυτή την κατανομή σε σχέση με αυτό το οποίο προτείνει ο Άντριου Νταφ και λαμβάνουν λιγότερες ή μεγαλύτερες η διαφορά είναι πολύ απλά πως ο συμβασμός του Cambridge ε, είναι γραμμικός και μετά πάνω κάνει ε, ένα τσάκισμα ενώ η δική μου η καμπύλη είναι πιο παραβολική. Πηγαίνει ομαλά σε όλο της ε, το μήκος και έχουμε άρα μια ευθύνη αναλογικότητα σε όλο το μήκος για να μην ε, έχουμε δηλαδή ένα τύπο τον οποίο να ακολουθούμε και στο τέλος να κάνουμε μια εξαίρεση και να μην το ε, ακολουθούμε. Μπορεί, έχετε και μια εικόνα μπροστά σας ε, τον πίνακα. Το αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας τύπος που βλέπετε πως στην αρχή ανεβαίνει απότομα και μετά γίνεται πιο ομαλός. Οπότε ε, βλέπετε πως υπάρχει αυτή η φθήνουσα αναλογικότητα και τα μεγαλύτερα κρατημέλη αναλογικά έχουν λιγότερες άρα έδρες. Και απορώ για το ότι ο Αντριοντάφ αναφέρθηκε στο γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο γιατί αυτό κατά την άποψή μου οδηγεί στο ότι θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις κατηγορίες ε, που ακούστηκαν περί μη ε, ισότητας ε, της ψήφου. Και αυτό βεβαίως θα πρέπει να γίνει με το να είναι όμοια η κατανομή σε όλες τις έδρες. Γι' αυτό έχω προτείνει αυτό το οποίο έχετε προτείνει. Βλέπετε και τις υπόλοιπες πληροφορίες πέρα από τον πίνακα. Ευχαρίστως να σας δώσω και άλλες ε, πληροφορίες. Υπολογίσαμε με 751, με 726, δηλαδή να έχουμε τις 726 συν 25 από μια πανευρωπαϊκή περιφέρεια και με δύο και με τρία επιπλέον κράτη-μέλη εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά ο τύπος. Ο τύπος λοιπόν τον οποίον ε, πρότεινα επίσης υπευλήθη στο Κέμπριτζ αλλά εκεί πέρα δεν έγινε δεκτός για λόγους που δεν μπορώ εγώ να κατανοήσω. Επίσης επειδή ο χρόνος πιέζει να πω κάτι άλλο. Προσωπικά θεωρώ πως εάν θέλουμε να το πάρουμε σοβαρά το θέμα με τους 25 βουλευτές από μια ενιαία ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια θα πρέπει να, για να γίνουν πιο ευρωπαϊκές οι ευρωεκλογέ, τότε οι 25 δεν θα πρέπει να προσθεθούν στην τωρινή κατανομή αλλά να συμπεριληφθούν στους 751 και τι θα γίνει έτσι δεν θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερο κοινοβούλιο γιατί βεβαίως θα μας πούνε θέλετε περισσότερα χρήματα, περισσότερες έντρες κτλ. Και δεύτερον δεν χρειάζεται να αλλάξει και η συνθήκη έτσι. Γιατί βεβαίω εκεί πέρα θα έχουμε αναγκαστικά αλλαγή της συνθήκης αν φύγουμε από τους 751. Να παραμείνουμε όμως σε αυτόν τον αριθμό δεν χρειάζεται. Συνολικά θα χαιρόμουν αν σε, τόσο, σε τέτοιες σκέψεις περί μεταρρυθμίσεων που αφορούν τους πάντες εδώ μέσα και την δημοκρατία να ε, συζητάμε περισσότερο μεταξύ μας από ό,τι έγινε μέχρι στιγμής και να επιλέγετε έτσι ο καλύτερος ε, τρόπος από το να προσπαθούμε να περάσουμε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε. Ε, κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω την, ε, τη βασική ιδέα, ευχαρίστως να συνεργαστώ, απλά απορώ για το ότι δεν αναζητήθηκε αυτή η συνεργασία. Νομίζω αυτό πρέπει να κάνουμε, εάν είναι να αλλάξουμε τίποτα έναντι και του Συμβουλίου. Δυστυχώς στις 10 έχουμε ψηφοφορία. Σας παρακαλώ να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Σαλάκο, ο οποίος είναι ο τελευταίος στον κατάλογο, να διακόψουμε τη συζήτηση για την έκθεση DAF, να ψηφίσουμε για την ε, έκθεση της κυρίας Γιαννάκου και κατόπιν μετά από την ψηφοφορία που ελπίζουμε ότι δεν θα κρατήσει πάρα πολύ ώρα, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για την έκθεση DAF. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σαλάτο και ελπίζω να είστε σύντομο. Πολύ σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η προσπάθεια που γίνεται εδώ για να δούμε του συνολικούς όρους για τη σύνθεση του επόμενου κοινοβουλίου προσπαθεί να εξυγχρονίσει και να ενοποιήσει τον τρόπο ε, έκφρασης ε, των κρατών μελών μέσω της ψήφου, των, της των πολιτών τους. Να σας πω καταρχάς ότι εμείς γνωρίζουμε στην Ευρώπη ότι υπάρχουν ε, χώρες μέλη που έχουν ε, ε καταλόγους, ε, λίστες με σειρά προτίμησης και ξέρουμε ότι υπάρχουν και κράτη-μέλη που ε, έχουν ψήφο με σταυρό προτίμησης. Ο κατάλογος, η λίστα, ε, ορισμένες φορές επιτρέπει στα κράτη-μέλη και στα πολιτικά κόμματα να επιλέγουν με βάση συμφέροντα. Σε χώρες όπως την Ιταλία, ο ο κατάλογος, η λίστα έτσι όπως είναι, δεν επιτρέπει στους ε, υποψηφίους ε, να ε, επιλέξουν και να φροντίσουν τους ε, πολίτες τους, ενώ επανεκλέγονται άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να εκλεγούν ακριβώς και μόνο γιατί βρίσκονται σε καλή θέση στη λίστα. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε και κάποια δυνατότητα ενοποίησης για τους ε, τρόπους με τους οποίους γίνονται οι εκλογές. Υπάρχει για παράδειγμα αυτό που υπενθύμισε ο συνάδελφος τη σημειανικτή λίστας. Ε, έτσι να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα όλοι. Επίσης η άλλη πρόταση που κάνω είναι να μην αγνοείται η γυναικεία παρουσία. Σε όλη αυτή τη διαδικασία αγνοείται η γυναικεία παρουσία. Μήπως θα έπρεπε να υποδείξουμε ε, στα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν σταυρό προτείνησης να υπάρχει και ε, ψήφος αναφύλων, δηλαδή να ψηφίζουν έναν άνδρα και μία γυναίκα του παραδείγματα. Ή στο άλλο εκλογικό σύστημα να υπάρχει μία ποσόστοση που θα αφορά τι γυναίκε ώστε και εμείς στην Ευρώπη να έχουμε την αίσθηση ότι σεβόμαστε το ρόλο και την αποτελεσματικότητα του ρόλου που διεξάγουν οι γυναίκες ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Όπως σας είπα, θα διακόψουμε τώρα τη συζήτηση για την έκθεση DAF, την οποία θα συνεχίσουμε αργότερα. Και θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία για τις ε, τροπολογίες για την έκθεση Γιαννάκου. Δεν ξέρω αν η κυρία Γιαννάκου θέλει να λάβει το λόγο πριν ε, ψηφίσουμε ή αν μπορούμε να ψηφίσουμε απευθεία. Παρακαλώ. Ε, Monsieur le Président, je fais deux, amendements de compromis encore. Έκανα δύο ακόμα συμβαστικές τροπολογίες και δέχτηκα και κάποιες παρατηρήσεις από κάποιους συναδέλφους. Έχουμε 12 τροπολογίες συμβιβαστικές και τις υπόλοιπες τροπολογίες οι οποίες ε, δεν ε, περιλαμβάνονται στη συμβιβαστική λύση. Σας παρακαλώ λοιπόν όταν θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε συμβιβαστικές τροπολογίες. Με να μας το πείτε για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη αυτές τις νέες συμβαστικές τροπολογίες, εντάξει. Λοιπόν, να ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 22, παράγραφος 1 του κυρίου Ντάφη. Υπέρ, ε, ανάταση χειρός παρακαλώ, όποιοι είστε υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23, από τον κύριο Ήλτσεφ. Υπέρ, Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Νταφ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Σέπφλιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Χάναν Van Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28 DAF. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29 29Τ, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρώτη συμβαστική τροπολογία τώρα η οποία καλύπτει τις τροπολογίες 30 και 32. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία υπέρ 36. Καταπίπτουν ε, οι 30 έως 35 και ψηφίζουμε τη 36. Σόλτς, υπέρ, Κατά. Απορρίπτεται. 11.9. Συμβαστική τροπολογία και πάλι εδώ που καλύπτει τις τροπολογίες 37, 38, 39 και 40. Στην παράγραφο 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επομένως, περνάμε στην συμβιβαστική τροπολογία D μετά από την τροπολογία 40 που καλύπτει τις τροπολογίες 41, 42, 43, 44, 45, 46 και 47. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 48 του κ για την 8β υπέρ, 8α συγγνώμη. Κατά. Έχουμε την ίδια πλειοψηφία με πριν, 11 ε, κατά 9 ε, υπέρ, επομένως απορρίπτεται. 49 και πάλι του κυρίου Χέφνερη. Υπέρ, Κατά. Απορρίπτεται. 10-10. Η τροπολογία 50 DAF υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51 της εισηγήτριας υπέρ. κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία. Εδώ έχουμε τρεις ε, τροπολογίες που μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού. 52, 53, 54 και η 55 είναι υπέρ της διαγραφής. Ε, ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν η τροπολογία υπέρ τη ε, διαγραφής και πάμε στην τροπολογία 55. Α, συγγνώμη, καταπίπτει λέει ο πρόεδρο. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία ε τη εισηγήτρια, η οποία καλύπτει τι 56, 57 και 58. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην 59, Ήλτσεφ. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία F που καλύπτει τις 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72 και 74. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Πρέπει να μετρήσουμε εδώ. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 75. Τροπολογία DAF. Συγγνώμη, διερθώνει ο Πρόεδρος. Στην 75, τον κύριο Χάναν, μία Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 76. Δαφ Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 77 και 78 ε, καταπίπτουν. Τροπολογία 79 του κυρίου Γκερέρο. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80 του κυρίου Νταφ και πάλι για διαγραφή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 81 Χέφνερ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 82 Λαμασούρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 83 Νταφ. Υπέρ. κατά εγκρίνεται τροπολογία 85 παράγραφος 23 και α, συγγνώμη συγγνώμη δεν ψηφίσαμε την 84 ήταν πάλι του κυρίου Νταφ και μπλέχτηκα τροπολογία 84 Νταφ λοιπόν υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 85 Γκρέτε Γκερέρο, υπέρ παρακαλώ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 86 Νταφ, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87 και πάλι την κυρίου Ντάφ, υπέρ διαγραφής. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 88, Γερέρο, υπέρ, <laughs> κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 89, υπέρ, Γιάννες Μπαρνεύο Γκαρθία, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 90 του κυρίου Γκλαφ Λάμστροφ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 91. Δαφ υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Γκουρμάι Γκερέρο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κύριε Γκουρμάη, μεγάλη επιτυχία. Κυρία Γκουρμάη, συγγνώμη. Τροπολογία 93 καταπίπτει, 94 επίσης. Τροπολογία 95 δάφ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Υπέρ, ξανά για να μετρήσουμε παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την επόμενη συμβαστική τροπολογία, συμβαστική τροπολογία G, που καλύπτει τις 97, 98, 99 και 96 υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία, συμβαστική τροπολογία και πάλι, α, που καλύπτει τις 1, 2, 3 8 και 17. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία υπερθμό 4 που είναι μια τεχνική διόρθωση. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ήλτσεφ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Γκραφ Λάμστροφ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 7. Σόλς υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία Γκουρμάη, τροπολογία 8 καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία Α, δεν την ψηφίζουμε. Τροπολογία 9 τη εισηγήτρια, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 12. Σόλτς. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 Έλτσεφ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 Χέφνερ. 13, συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος. Χέφνερ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται, λέει ο κύριος Μέντες Δεβίγο, εκτός μικροφώνου. 12-11 μετρήσαμε εμείς, λέει ο πρόεδρος. Ας κάνουμε μια επαλήθευση. Παρακαλώ όσοι δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν να μην ψηφίσουν. Κάποιος φωνάζει ότι δεν έχουμε κάρτες. Έχουμε κάποιους αναπληρωτές που ψηφίζουν χωρίς κάρτα. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω... Για κοιτάξτε πόσοι είναι εδώ από το ΕΛΚ. Νομίζω ότι είναι περισσότεροι από το, το, το νούμερο 9 το οποίο είπατε. Εννέα είναι η ψήφη του ΕΛΚ, τις έχουμε μετρήσει, αλλά τέλος πάντων να ξαναδοκιμάσουμε. Σας παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 13 Χέφνερ. Ανάταση χειρός. Δώδεκα. Κατά. 11 κατά. Επομένως, σωστά είχαμε μετρήσει. Για μία ψήφο εγκρίνεται. Τροπολογία 14, Χέφνερ, υπέρ. Ο κύριος Μέντες Δεβίου. Δεν είναι δυνατόν. Το ΕΛΚ είναι 9 και καταψηφίζουμε. Συν ο κύριος Σμιτ, ο κύριος Φόξ, ο κύριος Μπρόγκς. Δεν μπορούμε να είμαστε 11. Ο κύριος Μπρόγκς δεν υπερψήφισε. Τέλος πάντων, Είμαστε 12. 9, 10, 11. Α, καλά, δίκιο είχατε. Συγγνώμη, πρέπει να ξαναπάω στο δημοτικό. να μάθω να μετράω. Ε, δεν πειράζει, δεν κάνει κακό να επαληθεύουμε πότε πότε, λέει ο πρόεδρος. Ε, ξαναμετρήσαμε. Περνάμε. Θα πάω στο Cambridge, κύριε πρόεδρε, λέει ο κ. Μέντης Δεβίγο.

15 Χέφνερ υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Ε, Σήμερα, δηλαδή ξαναμπήκαμε τα κανονικά κωδικούς και το λέγαμε. Απορρίπτεται. 16 της κυρίας Γκουρμάη, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία Χέφνερ 17, που καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία Α, δεν ψηφίζουμε. Και η 18 καταπίπτει. 19, 20 και 21 που καλύπτουν τις τροπολογίες 19, 20 και 21 και ζητούν τη διαγραφή. Ο κύριος Μέντες Δεβίγο. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή καταψήφισε την παράγραφο 10. Επομένως, αφού καταψηφίσαμε την παράγραφο 10 και αυτό το, η αιτιολογική σκέψη αφορά την παράγραφο 10, ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να την ε, ε, ψηφίσουμε, γιατί καταψηφίσαμε την παράγραφο. Μισό λεπτό να το ελέγξουμε, λέει ο Πρόεδρος. Sí sequenza dovremmo votare anche qui nella stessa maniera. Dobbiamo votare però, o non si vota, o è decaduto. Si può, può dichiararlo caduto se vuole. Beh, mi pare che abbia ragione. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο συνάδελφος Μεντεστεβίγκο. Κύριε Ντάφ, ποιος είναι ο συνάδελφος Λόπεθ, τον είπε Λόπεθ τον κύριο Μεντεστεβίγκο, ο πρόεδρος. Κύριος Ντάφ, νομίζω ότι για να διευκρινίσουμε ότι είμαστε κατά του φορολογικού καθεστώτος για το προσωπικό του, των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων θα πρέπει να διαγράψουμε αυτή την αιτιολογική σκέψη ψηφίζοντας. Ο Πρόεδρος. Ούτως ή άλλως έχουμε συνοχή των όσων είπε ο κύριο Ντάφ, επειδή έχουμε ψηφίσει 10. Αν θέλετε να ψηφίσουμε απλώ για να το επαληθεύσουμε, ωραία. Ψηφίζουμε την αιτιολογική σκέψη ΑΑ που καλύπτει τι 19, 20 και 21. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Ωραία, εγκρίνεται. Η ούτω ή άλλω διαγραφή ζητάμε εδώ. Επομένω, ολοκληρώσαμε τι ε, τροπολογίε και μπορούμε να ψηφίσουμε το κείμενο όσο τροποποιήθηκε. Ποιο είναι υπέρ, παρακαλώ. Να, ψηφί... να μετρήσουμε αυτή τη φορά για να δούμε πόσοι είμαστε, παρόλο που είναι σαφή η πλειοψηφία. Κατά, μόνο μία ψήφος κατά. Ποιος, είναι, ε, ποιος απέχει? Α, συγγνώμη, δύο ψήφοι κατά, μία αποχή. Ωραία. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην κυρία Γιαννάκου. Παρακαλώ. Η κυρία Κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ κύριε Πρόεδρε θέλω απλώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, λέει κυρία Γιαννάκου, ε, από όλες τις πολιτικές πτέρυγες οι, οποίες, οι οποίοι με συνεπικούριζαν στην προσπάθεια και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά στην ε, Ολομέλεια όπως πήγανε και εδώ και ευχαριστώ. Να Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη δήλωση για την ψηφοφορία που μόλις έγινε. Και να ευχαριστήσω βεβαίως και την εισηγήτρια πάρα πολύ, ειδικά για τις ε, συμβαστικές τροπολογίες, τις οποίες ψηφίσαμε όλες πλην τις 10, όπου δεν συμφωνούμε με το σκεπτικό με συγχωρείτε, συμφωνούμε με το σκεπτικό, αλλά όχι με την ε, διατύπωση. Χτε ε, κατέθεσα μια δική μου πρόταση διατύπωση στην εισηγήτρια, την οποία θα καταθέσουμε ω προφορική τροπολογία στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να παρακαλέσω του συναδέλφου να το δουν προσεκτικά, γιατί δεν πρόκειται για ουσιαστική διαφορά, μόνο για διατύπωση, η οποία ξεκαθαρίζει κάτι το οποίο διαφορετικά θα ήταν ασαφέ και θα δημιουργούσε προβλήματα. Ε, ως πρόταση. Απλά να το δουν οι συνάδελφοι. Κατά τα λοιπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλό αποτέλεσμα και την ενσωμάτωση των διαφόρων θέσεων στην ε, τελική έκθεση. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση, αλλά στην ε, διαδικασία της ψηφοφορία. Είμαστε Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων. Γνωρίζω πως δεν συνηθίζεται να ψηφίσουμε εδώ πέρα, δεν συνηθίζεται να ψηφίζουμε με την κάρτα, αλλά καμιά φορά ε, μπορούμε για να διαπιστώσουμε ποιοι είναι από ποιες ομάδες να το κάνουμε ε, ηλεκτρονικά. Θα μπορούσε ο πρόεδρος να εξετάσει τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας. Γι' αυτό υπάρχει άλλωστε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, ο κύριος Γκέντς. Ευχαριστώ. Να επαναλάβω, χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι ψηφίσαμε με συντριπτική πλειοψηφία ε, υπέρ, αλλά χτες ε, μετά τη συζήτηση έδωσα, είπα πως ε, στη γραμματεία πως δεν ε, υπήρχαν στη συμβαστική λύση δύο τροπολογίες μου. Δεν αλλάζει τίποτα στο σύνολο, αλλά νομίζω πως ε, επειδή είμαστε και Επιτροπή Σταγματικών Θεμάτων θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ τυπικοί σε αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να μπορούμε να ενσωματώσουμε στις συμβαστικές τροπολογίες τις διάφορες απόψεις για να ψηφίζουμε έτσι ώστε είτε να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες ε, τροπολογίες για το περιεχόμενο τέτοιων ψηφισμάτων. Ωραία. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλες παρεμβάσεις για αυτή την έκθεση. Να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Γκουρμάη, λέει ο πρόεδρος. <laughs> Ποιος πρέπει να μιλήσει? Θέλει κάποιος το λόγο? Α, συγγνώμη. Τώρα μου εξήγησε ο γραμματέα. Την κυρία Γιαννάκου πρέπει να ευχαριστήσω. Οι ευχαριστίες λοιπόν έχουν ήδη γίνει και τώρα απλώ τις ε, ξαναδίνω θερμό στην κυρία Γιαννάκου για τη δουλειά που έκανε. Νομίζω ότι αναγνωρίστηκε και από του παρισταμένου, δεν χρειάζεται να πω και τίποτα περαιτέρω. Όσον αφορά τώρα την ηλεκτρονική ψηφοφορία, ειλικρινώ αν είχε κάποιο ζητήσει στη διάρκεια της ψηφοφορίας θα είχα πει ότι <coughs> μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν ε, αποφεύγουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί είμαστε συνταγματική επιτροπή. Απλώς ε, είναι πολύ πιο εύκολο να μετράμε με διανατάσσεω χειρός. Θα το λάβουμε υπόψη όμως. Ε. Να συνεχίσουμε τώρα τη συζήτηση για την έκθεση του συναδέλφου Νταφ για τον εκλογικό νόμο. Είχε ζητήσει το λόγο ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να επανέλθουμε σε αυτό που συζητούσαμε προηγουμένω ε, ε, ε, πριν αρχίσει αυτή η έκσταση που λέγεται ψηφοφορία. Οπότε σας παρακαλώ, δεν ξέρω αν είναι δυνατόν, αλλά συγκεντρωθείτε λίγο. Συνέδευε στην αίθουσα, ούτως ώστε ε, λίγο να έχουμε λίγη, λίγη ησυχία. Και σας παρακαλώ λέει ο πρόεδρος όποιος θέλει να φύγει να φύγει να μιλήσει έξω. Διότι το θέμα μας τώρα είναι σημαντικό. Caso quería volver al tema del voto preferencial. Quería volver al tema del voto preferencial. Όσον αφορά αυτή την ψήφο προτίμηση, με σταυρό προτίμηση τέλο πάντων, διότι είχε φανεί ότι υπάρχει συνένεση κατά, κατά της πρότασης για την ψήφο αυτή σταυρό προτίμησης, όμως άλλα ακούστηκαν μετά. Έχουμε διαφορετικές εμπειρίες, έχουμε την γερμανική εμπειρία, τελείως διαφορετική από τη δική μας, την ισπανική, διότι γίνεται αυτό στην γερουσία στη χώρα μου. Και ακριβώς το ίδιο κάνουν ε, και, και, ο λαός ε, ακολουθούν δηλαδή την κομματική γραμμή και ψήφισαν το ίδιο και για τη Βουλή και για την ε, Γερουσία. Το, πλεονέκτημα είναι ως επιτοπλίστων θεωρητικό. Το, το δε μειονέκτημα είναι κάτι το οποίο πρόκειψε στην πράξη η αρνητική εμπειρία από το Σταυρό Προτίμησης διότι πάρα πολύ συχνά αλλά όχι πάντα προξενεί εσωτερικές ε, προστριβές και υπάρχει ε, το ρίσκο του να έχουμε κάποιο είδους ε, αντικανονικές πληρωμές ή προβλήματα τέλο πάντων στις, στις εκταμιεύσεις για τους υποψηφίους. Οπότε τελικά οι ψηφοφόροι είναι δυνατόν να επιβληθούν και να έχουν την προτεραιότητα έναντι τη ιδεολογική πλατφόρμα του προηγούμενου προγράμματος των, ε, των κομμάτων. Πρόκειται επομένω για κάποια λίστα την οποία, η οποία έχει περάσει από κάποια διαπραγμάτευση μέσα στο κόμμα και έχει να κάνει με ιδεολογικέ αρχές. Όμως ε, υπάρχει και το θέμα του, του, του, του της μεταβλητής ε, της εθνικής κάτι το οποίο αλλοιώνει την, την βιολογική ταυτότητα, το ιδεολογικό προφίλ. Επομένως, γι' αυτό και στα το, βλέπουμε σαν πρόβλημα για τα κόμματα. Οι δε ε, οι ψηφοφόροι θα πρέπει να αποσυνδεθούν από το κόμμα, τον κομματικό μηχανισμό για να λειτουργήσει η δημοκρατία. Επομένως, για μένα είναι μεγάλο λάθος, λάθος ουσίας. Δεν έχουμε ε, την η δημοκρατία αν δεν είναι ισχυρά τα κόμματα, τα πολιτικά. Ούτε επίσης εδώ να έχουμε ευρωπαϊκή δημοκρατία αν δεν έχουμε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τα οποία να είναι επίσης αντίστοιχα ισχυρά. Και γι' αυτό εγώ λέω όχι στο, στην ψήφο με σταυρό προτίμηση γιατί νομίζω ότι στρεβλώνει την ουσία αυτού που θέλουμε ακριβώς να πετύχουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Γκερέρο και τώρα ο συνάδελφος Όντεγκαρντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την έκθεση. Και εγώ θα ήθελα να πω πως δεν θεωρώ πως ε, η πρόταση αυτή σημαίνει πως 16 ε, από τις 27 ε, χώρες θα χάσουν κάποιες έδρες και το εάν υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα υιοθέτηση. Εγώ θεωρώ πως ακολουθούμε το σωστό δρόμο εδώ πέρα όσον αφορά την ε, αναλογικότητα στην ε, σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο να εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες οι βουλευτές, αλλά βεβαίως δεν υπάρχει αναλογικότητα στο Συμβούλιο. Γι' αυτό είναι μονομερή συζήτηση, γιατί μιλάμε μόνο για μία πτυχή και όχι την άλλη, την σύνθεση δηλαδή του Συμβουλίου. Εάν το συγκρούν με, το ΙΠΑ που υπάρχουν δύο σώματα, εκεί πέρα υπάρχει αναλογικότητα όσον αφορά τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά στη Γερουσία κάθε πολιτεία, ανεξαρτήτως μεγέθους, έχει δύο γερουσιαστές. Έχουμε λοιπόν δύο σώματα ε, με ε, αναλογικότητα εμείς ε, εδώ πέρα και βεβαίως αυτό είναι απαραδεκτό δεν ξέρω δηλαδή αν είναι σωστό αυτό το οποίο είχε προταθεί αρχικά ότι δεν υπήρχε το εμπόδιο το κατόφλι του 5% όταν ε, φτιάχνονταν οι εκλογικές περιφέρειες. Όχι, πρέπει και αυτοί να εκπροσωπούνται, αλλά βεβαίως όταν μιλάμε για εθνική εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκεί πέρα το κατόφλι είναι πολύ υψηλότερο. Είναι 8%, 10% ή και 16%. Και θυμάμαι... Όταν η Τουρκία, θυμάστε, είχε βάλει ένα εκλογικό μέτρο 10%. Κάτι το οποίο θεωρήσαμε τελείως απαράδεκτο σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αλλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε εκλογικά μέτρα μέχρι και 16%. Γι' αυτό θεωρώ πως η πρόταση αυτή είναι περιορισμένη γιατί δεν λαμβάνει υπόψη ε, τις συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο. Γι' αυτό νομίζω πως θα πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω ακολουθώντας αυτό το οποίο έχει προτείνει ο Άντριου Ταφ. Ο κύριο Ταρκόφσκι. Very briefly... Uh, Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Τι γίνεται με κάποιον που μπορεί να είναι και δύο λίστε. Γιατί αυτό το συζητήσαμε, αλλά ε, το ζήταμε σαν δεχόμενο και δεν κατέβαινε τίποτα τροποπολογίες. Αν λοιπόν δεν θέλουμε να υπάρχει τέτοιου είδου διασυνοριακή ούτως ε, ναι. χρήση τη λίστα, του ψηφοδέλτιο, τότε κάποιο τι θα γίνει αν θέλει να πάει σε δύο ψυχοδέλτια. Γιατί εάν πούμε ότι κάποιο μπορεί να είναι εκεί, τότε θα είναι δύσκολο να πείσει κανεί ε, τα σπουδαία βαριά ονόματα που είναι στο κοινοβούλιο να θέλουν να πάνε σε αυτά τα ψηφοδέλτια. Αν όμω αφήσετε κάποιον, τότε υπάρχει πρόβλημα ότι ε, αυτού του είδου τα ψηφοδέλτια θα ε, θα πάνε σαν, σαν εθνικό ψηφοδελτίο. Οπότε... Τότε... Τότε κανεί εξετάζει πώ έχει πιο πιθανότητε να εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και απ' την άλλη, δεν έχει νόημα να συζητάμε για το μαθηματικό τύπο. Το έχετε σκεφτεί, Άντρου, ε, για πέστε μας, αυτό το πρόβλημα πώς προτείνεται να λυθεί. Yes, uh... Ο επόμενος, ναι. ναι. Η δημιουργία μιας υπερεθνικής περιφέρειας 25 ευρωβουλευτών ενώ προηγούμαστε οποιασδήποτε επιθυμίας του κοινού νομίζω πως θα γνωηθεί από τους ψηφοφόρους και θα καταλήξουμε σε τραγικά επίπεδα συμμετοχής στις εκλογές. Μας λένε πως οι υπερεθνικές αυτές λίστες θα ε, έχουν ισορροπία των δύο φύλων. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός ε, για εκλογικά συστήματα που προδιαγράφουν το αποτέλεσμα των εκλογών και το προφίλ των επιτυχημένων υποψηφίων. Εάν βεβαίως όλα τα άλλα ήταν ίσα, είναι πολύ επιθυμητό να έχουμε ισορροπία των δύο φύλων, αλλά και το τωρινό μας ποσοστό του 35% νομίζω συγκρίνεται με τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια του κόσμου. Το να λέμε στα κόμματα ποιον να επιλέψουν ως υποψήφιο και από πλευράς φίλου μοιάζει πάρα πολύ κοντά στο να <coughs> λέμε τι θα πρέπει να ψηφίσουν οι ψηφοφόροι καθώς περιορίζουμε τις επιλογές τους. Και το να λέμε στα φύλλα πως ε, το φύλλο είναι σημαντικότερο από όλα τα άλλα κριτήρια ενός υποψηφίου είναι παρέμβαση που πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μάλιστα επίθεση στο δικαίωμα των κομμάτων να αποφασίζουν ποιος ε, θα πρέπει να τους εκπροσωπεί και ποιος όχι. Λοιπόν, διάβασα την παράγραφο 2 της ε, έκθεσης του κυρίου Ντάφ και ελπίζω να μην παρεξήγησα. Λέει πως οι ψήφοι κατανέμονται είτε στην λίστα του κόμματος είτε σε συγκεκριμένους υποψηφίους εντός της λίστας. Εμένα αυτό μου φαίνεται πως ε, λέει πως θα μπορούν να επιλέγουν μετα, ε, εντός της λίστας οι υποψήφοι Δηλαδή μπορεί εγώ να βλέπω τη λίστα και να λέω «Α, εγώ θα τους βάλω στη σειρά που θέλω» ή να επιλέξω μια κλειστή λίστα. Καλά κατάλαβα, ναι. Αυτό έχει, ε, είναι πολύ θετικό για να, για να πω και κάτι θετικό. Ε, γιατί επιτρέπει στους ψηφοφόρους να, χωριστούν από μόνοι τους σε, μια, σε δύο διαφορετικές ομάδες, αν θέλετε, και θα μπορούν να περάσουν από τη μία ομάδα στην άλλη. Δηλαδή μπορούν να ξεκινήσουν να είναι έτσι λίγο πιο τεμπέληδες με την κλειστή λίστα και να περάσουν στην λίστα επιλογής. Και άρα τους επιτρέπει να αποφασίσουν μόνοι τους πόσο εξελιγμένοι θεωρούν ότι είναι. Αλλά δεν πρέπει να υποθέσουμε πως το να ενθαρρύνουμε την ατομική επιλογή στους ψηφοφόρους θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ισορροπία των φύλων η εθνοτική ισορροπία. Ε, γιατί αυτό βασίζεται στην υπόθεση πως ε, το, οι ψηφοφόροι είναι, ασχολούνται τόσο πολύ με αυτές τις ισορροπίες όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Μπρόντς και μετά Βιλάντερ. Ο κύριος Βιλάντερ. Ευχαριστώ. Η συζήτηση δείχνει πως δεν πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την έκθεση. Ε, δυσκολεύει πάρα πολύ η συζήτηση. Οπότε, ξεκινήσουμε από τις γυναίκες, ας πούμε. Σωστό και σημαντικό, αλλά αν δούμε πως σε 25 κράτη-μέλη στα εθνικά κοινοβούλια έχουμε λιγότερες γυναίκες, από ό,τι εδώ μέσα. Δηλαδή η Ισπανία έχει το ίδιο ποσοστό και στη Μάλτα είναι περισσότερες. Αλλά οι υπόλοιπες 25 χώρες έχουν λιγότερες. Αλλά δεν πρέπει να βάλουμε. Έχουμε πράγματα να κάνουμε, αλλά όχι ποσοστώσεις. Ε, ακούσαμε και τα διάφορα επιχειρήματα. Πρώτο. Δεύτερον, για τον ίδιο λόγο προσωπικά πιστεύω πως οι 25 αυτοί ε, βουλευτές είτε προστεθούν είτε όχι δεν θα πρέπει να πάνε σε εδώ πέρα την έκθεση. Μπορούμε να θέσουμε κάποια ζητήματα αρχής και μετά να δούμε ε, το τι θα γίνει. Δεν ε, θεωρώ... Είτε μπορούμε να τους ενσωματώσουμε στον τωρινό αριθμό, όπως πρότεινε ο κ. Σχέφνερ, αλλά δεν ξέρω, νομίζω μπορεί να χρειαστεί μια αλλαγή της ε, συνθήκης. Όσον αφορά τώρα το μέγεθος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μην ξεχνάτε πως είχε πει το Κοινοβούλιο πως ανεξαρτήτως διευρύνσεων εμείς θέλουμε 700 και το Συμβούλιο είχε μπει 750 ε, και μην ξεχνάτε οι υποδομές στο πέρα είχαν προγραμματιστεί για 700 μόνο τώρα για τις τροπολογίες οι οποίες κατέθεσα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες τροπολογίες, μια πρόταση για τον πληθυσμό. Κοιτάξτε, εγώ επέλεξα όμως την διατύπωση ο πληθυσμός της Ένωσης, που νομίζω είναι σωστότερη σκέψη. Μετά προσπάθησα να ορίσω πως 31 Δεκάτου αυτού του έτους να έχουμε πει πότε θα είναι οι εκλογές να τις έχουμε ορίσει για το 2014. Γιατί βεβαίως ε, εδώ πέρα μένουμε λίγο πίσω από τις προσδοκίες. Τώρα, τροπολογία 93. Παρατήρησα στο τέλος προηγούμενης θητείας πως κάποιοι επίτροποι παρετήθηκαν ε, έθεσαν υποψηφιότητα για βουλευτές, μετά προσπάσαν πάλι να γίνουν επίτροποι, κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι όχι. Εγώ θεωρώ πως καταραίει το σύστημα με το να απαγορεύουμε την υποψηφιότητα στους ε, επιτρόπους ε, ή στα μέλη της ΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών. Εάν θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκά πρόσωπα νομίζω καλό θα είναι να έχουμε αυτά τα άτομα στις ευρωεκλογέ για να έχουμε και μία λύση που θα αντέξει στο μέλλον κατόπιν ε, σας ευχαριστώ εδώ πέρα για αυτό το οποίο έχετε αναφέρει στην εκθεσή σας το ζήτημα της ασυλίας κατέθεσα αντροπολογία 108 για να αναφέρω μια περίπτωση που προέκυψε στο παρελθόν. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπου μπορεί όσον αφορά το δικαίωμα του εκλέγει να υποβληθούν κάποιες ε, αγωγές. Ε, έχει γίνει με την περίπτωση Ταπή, με την περίπτωση Λεπέν. Δεν νομίζω πως μπορούμε για αυτό ειδικά το ζήτημα, το δικαίωμα του εκλέγει να καταλήγουμε σε αγωγές και σε στικά δικαστήρια. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια λύση, αλλά αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι και μια λύση η οποία θα αντέχει και θα στέκει πολιτικά. Και μην ξεχνάτε πως εδώ πέρα κινδυνεύουμε με πολιτική αυτοκτονία στην ε, ε, Ήπειρο αυτή, γιατί κανείς δεν μπορεί, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εξηγήσει και να αντιληφθεί αυτούς τους τύπους και τις πολιτικές φόρμουλες. Θα πρέπει να μπορούμε να το εξηγήσουμε σε ένα 17χρονο μαθητή το τι συμβαίνει και να το καταλάβει και να μπορεί να το εξηγήσει ας πούμε στην τάξη του στο σχολείο και αυτός. Γιατί απομακρυνόμαστε όλο και ε, περισσότερο από τον λαό που υποτίθεται ότι εκπροσωπούμε. Γι' αυτό έχω άλλη μια πρόταση. Με κάθε σεβασμό για τους συναδέλφους εδώ πέρα, τον κύριο Ράγγελ και τους λοιπούς, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Νταφ ε, με τις ε, νομικές κατηγορίες του Ομοσπονδιακού Γερμανικού Δικαστηρίου. Δεν είναι θέμα μια χώρα που έχει 96 βουλευτές έχει πρόβλημα να χάσει κάτι. Αν το πάρουμε τελείως αναλογικά, η Γερμανία έπρεπε να έχει 130 και η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία πάνω από 100. Οπότε, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη διόρθωση προς όφελος των μικρότερων χωρών. Οπότε το θέμα μας δεν είναι να κακομεταχειριστούμε τους μικρούς, είναι να έχουμε ένα, μια λύση η οποία θα αντέξει στα δικαστήρια και θα εφαρμόζει την ευθύνουσα αναλογικότητα. Πριν γίνω νομικός και δικηγόρος ήθελα να σπουδάσω μαθηματικά και ε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής. Ε, δεν μπορούμε να πούμε πως ε, τηρείται η φθήνουσα αναλογικότητα αλλά στην τελευταία έδρα κάνω μία εξαίρεση. Θα πρέπει με μία κάποια νομική, ε, μαθηματική με να υπάρχει μια α, παραβίαση αν θέλετε της αναλογικότητας αυτής δεν θα πρέπει λοιπόν να δίνουμε την εντύπωση πως με μια πολιτική φόρμουλα πως κάνουμε κάποια παζάρια εδώ πέρα θα πρέπει να έχουμε συστήματα τα οποία θα είναι λογικά και θυμάμαστε τι είχε γίνει αυτό με την έκθεση Λαμασούρ Σεβερίν στο σώμα Και βεβαίως, εντάξει, υπάρχει η αρχή μία ψήφο ανά άτομο, αλλά έχουμε τις έξι έδρες που είναι το μίνιμουμ. Οι υπόλοιπε μετά κατανέμονται ε, σύμφωνα με το σύστημα DEONT και όταν φτάσουμε στο νούμερο 90 έχουμε ένα πλαφόν και μία ανακατανομή των υπολείπων. Είναι ένας ε, αυτοματισμός που ενισχύει τις μεσαίες χώρες και πλην ε, τεσσάρων περιπτώσεων δεν αποκλίνει από την τύπο του κυρίου Νταφ. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η Πορτογαλία θα έχει μία παραπάνω έδρα, η Πολωνία μία παραπάνω έδρα, η Γαλλία και η Ισπανία θα έχαναν από μία, αλλά είναι ένας αυτοματισμός που θα ισχύσει και για το μέλλον. Γιατί εάν είναι πολύ λεπτομερής ο τύπος θα πρέπει κάθε φορά να εισάγουμε νέα κριτήρια για να λειτουργήσει και είναι δύσκολος μηχανισμός. Οπότε εγώ θεωρώ 6 συντεόντ και πλησιάζουμε ε, σε αυτό το οποίο τώρα προσπαθούμε να επιτύχουμε με πάρα πολύ δύσκολους τύπους. Ο Deont είναι πολύ απλό σύστημα η διαφορά εδώ πέρα είναι πως με τα μικρά νούμερα, δηλαδή αν έχουμε 700 άτομα και πρέπει να έχουμε μια επιτροπή με 18, εκεί πέρα υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αλλά με μεγάλα νούμερα, στους 750, οι διαφορές είναι ελάχιστες. Όλα τα συστήματα είναι κάπως γραμμικά. και οι διαταραχές είναι μικρές. Γιατί μην ξεχνάτε, ο κύριος Ντεόντ δεν είναι κανένας τυχαίος μαθηματικός από το Κέμπριτζ. Ε, γύρισε όλες τις, ε, τις επιτροπές, ε, όλο το κοινοβούλιο. Τον εκτιμούν όλοι, είναι γνωστός. Δεν υπάρχει λόγος έτσι να τον απορρίψουμε Χωρίς δεύτερη σκέψη. Um Συγγνώμη. Και αν ε, ορίσουμε αυτή την αρχή, κύριε Νταφ, τότε συμφωνώ μαζί σας για να αποφύγουμε τη μεγάλη αλλαγή. Αν πούμε τώρα πως ορίζουμε την αρχή για το 2019 και δάνουμε τη σημερινή κατάσταση φτάσουμε σε ένα συμβασμό το 2014 και το 2019 θα εφαρμόσουμε την αρχή την οποία αναφέρουμε σήμερα. Και μην ξεχνάτε, ο, ο πληθυσμός που ορίζεται ως κριτήριο. Στο τέλος αυτού του έτους πρέπει να είναι γνωστό το νούμερο, έτσι ώστε τέλος του 2012 να έχει ε, υπολογιστεί ο αριθμός των ε, βουλευτών. Αλλιώς ε, θα έχουμε αργήσει πάρα πολύ και μετά θα έχουμε Ευχαριστώ Ευχαριστούμε τον κύριο Βίλαντ. Ο κύριο Σάντερκαρ τώρα. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλύτερα να σας τα πω αγγλικά για να σας τα πω καλύτερα. Είναι μεγάλη μου χαρά που βέβαια έχουμε του διερμηνία, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι το θέμα είναι απλούστερο από ό,τι φαίνεται από τη μαθηματική φόρμουλα. Έχουμε κάποιους καθηγητές του Cambridge, οι οποίοι νομίζω ότι είναι 100% ε, σωστοί σε αυτό το οποίο λένε. Όμως το ερώτημα το οποίο τους τίθεται έχει διατυπωθεί λάθος. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί αυτό το οποίο μας ε, λένε τώρα είναι μια γραμμική αναλογικότητα. Ε, γιατί να μην θεωρηθεί απόδεκτη πρόταση. Όμως η ουσία είναι ότι αυτού του είδους η ορολογία φθήνους αναλογικότητα σημαίνει μη γραμμική αναλογικότητα. δεν σημαίνει έξι έδρες για αυτούς που θα είχαν μηδέν. Δηλαδή, για, τα, για τις μικρότερες χώρες υπάρχει περισσότερη εύνοια από το σύστημα παρά από, για τις μεγαλύτερες χώρες. καλύτερα οι μικρές παρά οι μεσαίες χώρες και για τις πιο μεγάλες ακόμα λιγότερο ευνοϊκό το σύστημα. Πολύ απλό είναι. Και επομένως αυτό θα μπορούσε να γίνει. Είναι όμως μη γραμμικό, όπως το είπε ο συνάδελφο Χέφνερ. Άρα, αυτού του είδου η προσέγγιση είναι μοναδική. Υπάρχουν παράμετροι, υπάρχουν πολλέ παραλλαγέ λαμβάνοντας και υπόψη γίνεται στη Γερμανία. Αλλά η ουσία των πραγματών ποια είναι. Δεν ξέρω, γιατί δεν ήμουν στις διαπραγματεύσεις. Ο Λαμασούρ και ο Σέβερν δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν, αλλά η κατάληξη των διαπραγματεύσεων είναι αυτό, αυτή η πρόταση που όμως δεν είναι γραμμική. Έτσι εκ των τον το βγάλαν αυτό. Πώς έγινε. Μπορεί κανείς να φτιάξει μια γραφική παράσταση, αλλά αυτό εδώ είναι αλλιώ, είναι, είναι γραμμικό, είναι ευθύγραμμο. Άρα λάθο ετέθη ε, η, το, ερώτημα στου καθηγητέ. Το, το DP2 ήταν λάθο. έχουμε δύο χώρε πάρα πολύ κοντά που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό και μετά δίνουμε μια, ένα έδρανο παραπάνω στη μία από τις δύο, όμως αυτό είναι ασυνεπές. Είναι άδικο. Οπότε οι μαθηματικοί διαστρέβλωσαν το, τη γενική αρχή της, ε, της, της γραμμικής αναλογικότητας. Πάρα πολύ απλό. Γίνονται αυτά όμως. Γίνονται συχνά. Άρα, καλή αυτή η μαθηματική, αλλά του ετέθη λάθος το θέμα. Το θυμάμαι αυτό, γιατί πριν από 20 χρόνια είχα ασχοληθεί με τα μαθηματικά, σε, τα εφαρμοσμένα, στη βιολογία κλπ. Άρα το θέμα είναι πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις, αυτές οι ιδέες κάποιων που προέρχονται από άλλο για να το καταλάβουν οι μαθηματικοί, οπότε οι μαθηματικοί μετά να μπορούν να διεκπεριώσουν το πρόβλημα, το λύσουν. Άρα, εάν τώρα πούμε ότι φεύγουμε από την φθήνουσα αναλογικότητα και όλες οι χώρες θα υπαχθούν σε αυτή την, την γραμμική ε, αναλογικότητα θα έχουμε αυτή την περικοπή το κόψιμο αυτό πάνω και κάτω χάνει η Λιθουανία εγώ σαν πολιτικός Πρόκειται να προστατεύσω τα συμφέροντα της χώρας μου και θα εξηγήσω ότι παραβιάζεται το γράμμα και το πνεύμα της νίκης της Λισαβόνας. The last point, of course, is uh, because that... Τώρα το τελευταίο. So I, I cannot... Και ο Γιαγέλα τελικά με συμβασμό έφυγε από τη Λιθουανία, πήγε στην Πολωνία, έγινε Βασιλιά, επομένω, δεν, δεν, φταίει, δεν η μαθηματική. Ήρθε αντιπρόεδρο ο Επίτροπο Εύκοβιτ, τον οποίο ζητώ συγγνώμη πριν του δώσω το λόγο, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο και τη μεταρρύθμιση του. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντάφ, λοιπόν, για να απαντήσει στις πολύ άριθμες παρεμβάσεις ε, που ακούσαμε ε, πριν από λίγο. Κύριε Ντάφ. Ε, Εγώ περιμένω από τον Επίτροπο ενδιαφέρον έντονο για το θέμα το οποίο συζητούμε. Γιατί έχει σημασία πολιτική και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε δίκιο όλοι όσοι ανέφεραν ότι επειδή ψάχνουμε ένα μαθηματικό τύπο για την κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο δεν ελάβαμε υπόψη την εκπροσώπηση των χωρών στο Συμβούλιο. Όμως αυτό δεν είναι στην εντολή μας. Ελπίζω ότι η Λισαβόνα θα το ρυθμίσει το ζήτημα αυτό όσον αφορά το Συμβούλιο. Τουλάχιστον στο ορατό, στο προβλέψιμο μέλλον. Έχουμε δει τι διαδρομέ έχουν γίνει όσον αφορά τι μεταβολέ στην σύνδεση του Κοινοβουλίου τελευταία δεκαετία και να δούμε κατά πόσον μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη για τη σύνδεση του Κοινοβουλίου και να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε μια ε, άνοδο, μια ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας που μας περιβάλλει. Νομίζω ότι κάπω έτσι. Αυτά ήταν τα κίνητρα τέλο πάντων των όσων ε, προσπάθησαν κάτι να πετύχουν. Φυσικά και κάποιοι ανέφεραν ότι δεν υπάρχει 100% στεγανό μαθηματικό σύστημα. Αλλά στην εντολή μας περιέχεται το ότι θα πρέπει να κινούμε θα γίνεται πιο επιστημονικά και έτσι να αντισταθμίζουμε κατά κάποιο τρόπο να είμαστε αντίβαρο στην κομματοκρατία του, του, του, του κόμματος από το οποίο προερχόμαστε. αυτά συμφωνήσαμε και τα είπαμε στους ε, μαθηματικούς. Δεν θεωρώ ότι έγινε επί βάσης αυθαίρετης αυτός ο συλλογισμός. από τους ε, πανεπιστημιακούς του Cambridge. Γιατί φυσικά έχουν στέρεα θεμέλια πανεπιστημιακά, ακαδημαϊκά αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι βάσιμες αυτές οι επικρίσεις του. Ότι πήγαμε σε κάποιους οι οποίοι θα μεροληπτούσαν κλπ. Αυτό νομίζω είναι προσβλητικό σε σχέση με την φήμη τους αλλά και την εγκαιρότητά μας. Το βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει τώρα να μας απασχολήσει όμως είναι το εξής. κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε σαν κοινοβούλιο σύμφωνα με τα οποία σύμφωνα με όσα προβλέπει συνθήκη. Μπορούμε να τα αφήσουμε στο Συμβούλιο και εμείς να ελιχθούμε όσο γίνεται σε πολιτικό επίπεδο στις διαπραγματεύσεις. Εγώ Πάντω νομίζω ότι είναι καλύτερα να ακολουθήσουμε αυτό το μαθηματικό τύπο στι διαπραγματεύσει. Καλά, να λάβουμε υπόψη τι προτάσεις όπως έχουν υποβληθεί. Αλλά θα πρέπει και αυτοί που διατύπωσαν αυτέ τι προτάσεις θα πρέπει να τις τεκμηριώσουν όσο γίνεται πληρέστερα. Τώρα, λοιπόν, όσον αφορά τα ψηφοδέλτια να είναι ανοιχτά ή να είναι εν μέρει ανοιχτά, Εγώ συνεχίζω και θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει την επιλογή ο πολίτης έχετε δηλαδή μια, ένα ψηφοδέλτιο, μια λίστα που να είναι καθορισμένη αυστηρά από το κόμμα ή να μπορεί να διαλέξει ένα συγκεκριμένο υποψήφιο. Νομίζω ότι είναι καλύτερο. Έτσι νομίζω ότι ισχύει πέσοντες δημοκρατίες. Φυσικά και προτιμώ να είναι τα κόμματα ισχυρά. Αλλά από την αρχή αυτής της θητείας ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να εδρεωθούν, να αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία και κύρος αυτά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, κάτι και το οποίο νομίζω συμβαίνει. Όμως τώρα, ε, κατά κάποιο τρόπο είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζουμε το να κάνουν κάτι ουσιαστικό αυτά τα κόμματα και οπότε άρα να προσέξουμε να μην υπερβάλλουμε στον αφορά το πόση ισχύ θα έχουν αυτά τα κόμματα. Τώρα το άλλο ερώτημα ήταν το αν μπορεί κάποιος υποψήφιος να είναι και σε υπερεθνική και σε εθνική λίστα ψηφοδέλτιο τέλο πάντων. Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, εγώ απαντώ ναι, διότι έτσι δίνεται κίνητρο στον κόσμο να πάει και στην υπερεθνική λίστα, στο υπερεθνικό ψηφοδέλτιο. σε κάποιες χώρες Βέβαια, θεωρείται σκανδαλώδες το να βρίσκεται κανείς σε δύο ψηφοδέλτια. Καλά, θα μπορούσε να ληφθεί απόφαση με κάποια ψηφοφορία. Θα δούμε. Αυτό το αποφασίσουμε άπαξ και το σκεφτούν όλοι. Ο Μπρόξ είπε ότι θα έχουμε μεγάλη αποχή. Ε, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοινική η αντιμετώπιση που γίνεται για τα εθνικά πολιτικά κόμματα. όσον αφορά την ε, πλατφόρμα των προτάσεων τους για την Ευρώπη. Οι εκλογέ έχουν εθνικό χαρακτήρα. Καμιά φορά και εθνικιστικό. Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα. Πάρα πολλοί ψηφοφόροι θα ήθελα να έχουν αλλιώς τα πράγματα. Θα ήθελα να δει κάποιο είδου ομοσπονδιακό χαρακτήρα να έχουν τα πολιτικά κόμματα. Και έτσι να αντιμετωπίζονται αντίστοιχα και τα θέματα τα οποία απασχολούν τα κόμματα. Θα δούμε, θα δείξει. Πάντως και άλλα αξιόλογα ελέγχθησαν κ. Βίλαντ επίσης εξήγησε αυτά τα οποία έχει προτείνει και θα τα μελετήσω προσεκτικά. Και όπως προείπα, θα κανονίσω μια σάντηση με τους σκιώδεις ηγητές και εκεί μπορεί να έρθει όποιος άλλος ενδιαφέρεται. Και μπορεί να προτείνει ό,τι θέλει. Την επόμενη τρίτη. Ελπίζω θα συμφωνήσουμε και ότι θα κάνουμε κάποια εκτέλεση συνεδρία στην Επιτροπή μας ε, στις 7 ε, του μηνός στο Στρασβούργο. Οπότε θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νταφ και γιατί το καθήκον που έχετε να λάβει είναι ιδιαίτερα σκληρό. Προσπαθείτε να συμφωνήσουν όλοι και να καταλήξουμε σε θετικό συμπέρασμα ε, για τον εκλογικό νόμο. Αυτό που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα Εθνικά Κοινοβούλια, πολλό δε μάλλον και για τα ε, Ευρωκοινοβούλια. Να σας κάνω κι εγώ μια παρατήρηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο βασικών τάσεων που είναι εμφανή σε όλη την ευρωπαϊκή διαδικασία η τάση που είναι ε, να έχουμε απλώς ε, ένα υπερεθνικό χαρακτήρα και η τάση της ολοκλήρωσης. Επειδή όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι η έκφραση των λαών και θα πρέπει ε, στο τέλος να είναι με αναλογικό τρόπο η εκπροσώπηση, η εκλογής αντιλαμβάνονται μεν ότι υπάρχουν όρια, αλλά υπάρχει και η ανάγκη να υπάρχει και μια κρατική παρουσία, όπως γίνεται στο Συμβούλιο. Είναι λογικό λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν αυτές οι δύο τάσεις, επομένως πρέπει να βρούμε μια μέση εδώ. Και νομίζω ότι ε, είναι απλό αυτό που υπόθηκε, ότι θα καθορίσουμε έναν τρόπο εκπροσώπησης και για τις μικρότερες χώρες, <coughs> που σημαίνει ότι θα γίνει μια θυσία και για τι μεγαλύτερε χώρε, και έτσι θα προχωρήσουμε με αναλογικό τρόπο από εκεί και πέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα. Η απέτηση να δίνουμε υπερβάλλον βάρος ε, στα κράτη είναι μια απέτηση που ε, ε, πόρο απέχει από την ολοκλήρωση κατά την άποψή μου. Θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Ευχαριστώ κύριε Νταφ. Ε, και τώρα είναι εδώ ο Επίτροπος Σεύκοβιτς και θα πρέπει να δούμε τα σημεία 10, 11 και 12 στην ημερήσια διάταξη που αφορούν την τροποποίηση του κανονισμού για τις ακροάσεις των επιτρόπων. Και πάλι ο κύριος Ντάφη είναι ο εισηγητής για το σημείο αυτό και ε, έχουμε διαρθρώσει και διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, όσον αφορά το θέμα των ε, της ακροάσεων των οριστών των επιτρόπων ακούσαμε μια πρώτη παρουσίαση και συζητήσαμε και 12 τροπολογίες ε, τον Ιανουάριο, αλλά βάσει και τη συμφωνία πλαίσιο η Επιτροπή μας θα πρέπει να ε, διαβουλευτεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση τροποποίηση του κανονισμού. Γι' αυτό ακριβώς είναι εδώ ο Αντιπρόεδρος ε, Σεύκοβιτς, στον οποίο θα ήθελα να δώσω το λόγο για να μας πει την άποψή του για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Λέει ο κύριος Νταφ. Ε, ξέρω πως με έχετε βαρεθεί σήμερα το πρωί. Αλλά θα ήθελα να παρουσιάσω τις προτάσεις και μια αλλαγή που έκανα σε αυτές πριν ε, μιλήσει ο Επίτροπος. Νομίζω πως θα διευκολύνει την κατάσταση. Ε, με την άδεια του Επιτροπού, ο οποίος ο Επιτροπός δεν με άκουγε εξάλλου από το πρωί. Η συμφωνία πλαίσιο υποχρεώνει την ε, Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν στην ε, διαδικασία των ακροάσεων και στην διαδικασία έγκρισης ε, των επιτρόπων. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα διαβούλευσης, πρέπει να συμφωνήσουμε εμείς με την Κομισιόν. Και η αρχική μου πρόταση συμπεριελάμβανε την καινοτομία του ότι απαιτούσε από τον εκλεγμένο πρόεδρο της Κομισιόν να έρθει ενώπιον του Κοινοβουλίου και να εξηγήσει την κατανομή των χαρτοφυλακίων. Νομίζω πως ε, αυτό έλειψε στις προηγούμενες ε, ακροάσεις και το Κοινοβούλιο δεν ε, αντιλαμβανόταν ε, τις αποφάσεις του Προέδρου όσον αφορά την κατανομή των χαρτοφυλακίων και ήταν έλλειψη από πλευράς Κοινοβουλίου έπρεπε εμείς να επιμείνουμε αλλά θεωρώ επίσης πως η διαδικασία των ακροάσεων των επιτρόπων έγινε πιο προβληματική. Λόγω του ότι ε, δεν συζητήσαμε με τον πρόεδρο Μπαρόζο την απόφασή του για την σύσταση του σώματος ε, των επιτρόπων. Οπότε είχα προτείνει να προσκαλέσουμε τον εκλεγμένο πρόεδρο της Κομισιόν σε μια κοινή συνεδρίαση των, ε, της διάσκεψης των Προέδρων και των Προέδρων των Επιτροπών. Ο κύριος Μπαρόζο μου επισήμανε πως εάν υποχρεωθεί να δώσει εξηγήσει στο κοινοβούλιο για τις αποφάσεις του για τα χαρτοφυλάκια θα υποχρεωθεί να κάνει το ίδιο και ενώπιον του Συμβουλίου και αναγνωρίζω πως είναι πολύ σημαντικό μέρος ε, της ε, εξουσίας του εκλεγμένου Προέδρου το ότι λαμβάνει την απόφαση αυτός ή αυτή για την κατανομή των χαρτοφυλακίων. Εάν το Κοινοβούλιο κατά λάθο ε, μείωνε τον ε, ρόλο του εκλεγμένου πρόεδρου θα ήταν κάτι το λανθασμένο. Οπότε απέσυρα την ε, τροπολογία 1 υπάρχει μόνο και αντευτής ε, θα καταθέσω στο ψήφισμα και όχι στην διαδικασία που θα ε, συνοδεύσει την αλλαγή αυτή μία παράγραφο την οποία έχω μοιράσει. που σημειώνει απλά πως ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί, έχει την δυνατότητα να προσκαλέσει τον εκλεγμένο πρόεδρο της ε, Κομισιόν ε, για να ημερώσει το Κοινοβούλιο για την κατανομή των χαρτοφυλακίων. Και ελπίζω ο Επίτροπος, ο κ. Σεύσεβιτς, να μπορεί να μας διαβεβαιώσει πως ε, με την αλλαγή αυτή θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσει του Πρόεδρου Μπαρόσο και των διαδόχων του. Αυτά θα ήθελα να αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να ακούσω τι έχει να πει η Κομισιόν. Ευχαριστούμε κύριε Νταφ. Πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο, θα ήθελα να προτείνω να συζητήσουμε τα σημεία 11 και 12, να ζητήσω δηλαδή από τον Επίτροπο να μας τα παρουσιάσει και τα δύο από κοινού, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον ο κανονισμός αυτός ε, και η τροποποίησή του σχετικά με τις ακροάσεις των οριστών επιτρόπων ε, και το θέμα του διαρθρωμένου διαλόγου είναι εξίσου ενδιαφέρον αλλά δεν έχουμε και μεγάλες νομοθετικές αρμοδιότητες. Παρακαλώ λοιπόν κύριε Επίτροπε μπορείτε αν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει να συζητήσετε και τα δύο θέματα μαζί για να περιορίσουμε και το χρόνο και να αφήσουμε περισσότερο χρόνο για συζήτηση γιατί έχουμε και καθυστερήσει λίγο σήμερα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω λοιπόν να παρουσιάσω και τα δύο θέματα ταυτόχρονα για να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω το θέμα αυτό το οποίο παρουσιάζεται τόσο εύγλωτα στην έκθεση του κυρίου Νταφ. Η έκθεση για τις ακροάσεις των οριστέντων επιτρόπων και η πρόταση που γίνεται στην έκθεση αυτή ε, για αλλαγές ε, στον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας συγχαρώ. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά με αυτή την έκθεση. Έχετε μελετήσει προσεκτικά την όλη διαδικασία των ακροάσεων που έγιναν ε, και στην Επιτροπή σας. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, θα ήθελα να πω ότι στις περισσότερες παρουσιάσεις και στα περισσότερα σημεία της έκθεσης ε, ε, θεωρούμε ότι έχουμε βελτιώσει σε σχέση με τις ακρεάσεις και τον τρόπο που διεξάγονταν στο παρελθόν. Ε, χαιρετίζω και την προφορική τροπολογία που έκανε ο κύριος Ντάφ εδώ στην Επιτροπή γιατί νομίζω ότι έτσι διαγράφουμε το προφανές θεσμικό πρόβλημα που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι με τις αρχικές προτάσεις θεωρούσαμε ότι γίνεται παραβίαση της θεσμικής ισορροπίας και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όπως κατανέμονται μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προφορική τροπολογία λοιπόν του κυρίου Νταφ ε, βρίσκει σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι λαμβάνει υπόψη και την τρέχουσα θεσμική ισορροπία, τη συνθήκη της Λισαβόνας και επιπλέον ε, βρίσκει και έναν τρόπο να αυξήσει αυτό που ζητούσε ο κύριος Ντάφ, καλύτερη διαφάνεια και να κατανοούν καλύτερα οι Ευρωπαίοι πολίτες γιατί ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτός που καθορίζει τα χαρτοφυλάκια των επιτρόπων ε, κατά το συγκεκριμένο τρόπο και γιατί επιλέγει ε, τους ε, ανθρώπους που επιλέγει για τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο έλειπε από την ε, προηγούμενη διαδικασία και νομίζω ότι ο κύριος Νταφ δίνει τη δυνατότητα πλέον ε, να αυξηθεί η διαφάνεια για την όλη διαδικασία και να κατανοήσουν καλύτερα οι Ευρωπαίοι πολίτες πώς γίνεται η κατανομή, η ε, ανάθεση των χαρτοφυλακίων και οι συγκεκριμένοι διορισμοί των επιτρόπων για να διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Τώρα, κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες στην έκθεση του κυρίου Νταφ. Χαίρομαι που μπορούμε να το συζητήσουμε, διότι όπως είπε και ο πρόεδρος, αυτή η διαδικασία περιλαμβάνεται σε συμφωνία πλαίσιο. Έτσι μπορούμε και εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεμβαίνουμε επί, τα θέματα, ε, επί των θεμάτων αυτών και άλλωστε αυτά τα θέματα αφορούν του επιτρόπου. Κάποιο που έχει περάσει μια διαδικασία ακρόαση γνωρίζει πόσο σημαντική είναι και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε σαφεί και διάφανου κανόνε. Είμαστε υπέρ τη τάση λοιπόν που προτείνει ο κύριο Νταφ στην ε, έκθεσή του όπου ζητά να υπάρχουν σαφείς, ε, διάφανοι, οριζόντιοι κανόνες για κάθε ένα από τα στάδια των ε, κοινοβουλευτικών ακροάσεων. Γνωρίζουμε ότι χρειάστηκε να ε, αυτοσχεδιάσουμε σε κάποιες περιπτώσεις το παρελθόν. Νομίζω ότι στην πολιτική είναι δύσκολο να αποφύγουμε τους αυτοσχεδιασμούς στο 100% αλλά όσο πιο ε, σαφείς και πιο οριζόντους κανόνες έχουμε τόσο πιο διάφανη είναι η διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο σε αυτές τις ε, οριζόντιες διευθετήσεις, κυρίως όσον αφορά τη διάρθρωση της ακρόασης, την αξιολόγηση και φυσικά θα θέλαμε να υπήρχαν και ελάχιστες πτυχές οι οποίες θα αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια τη κάθε επιτροπής. Τι εννοώ με αυτά τα σχόλια. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα ήταν θετικά θετικό θα ήταν να έχουμε ένα κανόνα ο οποίος θα δίνει τον ίδιο χρόνο για κάθε ακρόαση. Διότι Αυτό θα ενισχύσει την οριζόντια ε, προσέγγιση και την ισότιμη μεταχείριση για όλους τους επιτρόπους που έρχονται σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πες, ε, δεύτερο σημείο, θεωρώ ότι ο καθένας από τους οριστές της επιτρόπους θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να κάνει μια αρχική παρέμβαση, παρουσίαση και να ε, ε, πει κάποια πράγματα για τις προτεραιότητές του ή τις προτεραιότητές της πριν ξεκινήσει η συζήτηση με ερωταποκρίσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και ε, τη διάρκεια των εισαγωγικών παρεμβάσεων είχαμε ξεκινήσει με 20 λεπτά, μετά το περιορίσαμε στα 10 λεπτά. Εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θεωρούμε ότι δεν είναι εύκολο να παρουσιάσει κάποιος όλες του τις προτεραιότητες και όλες του τις δεσμεύσεις εντός 10 λεπτών. Ε, εάν βέβαια είναι η απόφασή σας αυτή θα τη σεβαστούμε. Ε, σας ζητώ όμως να το ξανασκεφτείτε μήπως τα 10 λεπτά είναι... λίγος χρόνος, διότι ξέρουμε ότι μία αρχή, ακροάση διαρκεί περίπου τρεις ώρες. Τώρα και κάποιε επιπλέον διαδικαστικές πτυχές των ακροάσεων. Γνωρίζετε ότι όλη αυτή η διαδικασία ξεκινά με ένα ερωτηματολόγιο. Θεωρώ λοιπόν εδώ ότι καλό θα ήταν ο κάθε επίτροπο να έχει τη δυνατότητα να σχολιάσει ίσο αριθμό προτεραιοτήτων της Επιτροπής και θα πρέπει να βρίσκονται και στο πεδίο εφαρμογής του χαρτοφυλακίου του. Όσον αφορά τώρα την όλη διαδικασία και για να υπάρχει καλύτερη οριζόντια αξιολόγηση των ακροάσεων στη συνέχεια και καλύτερη προετοιμασία των επιτροπών για τη συζήτηση, αν ε, ε, γίνει, καλό θα ήταν να ομαδοποιούνται οι ερωτήσεις αναθεματικές κατηγορίες. Αυτά όσον αφορά την προετοιμασία για τις ακροάσεις, τα ερωτηματολόγια και τις ακροάσεις αυτές καθεαυτές. Τώρα, περνάμε στη φάση μετά την ακρόαση, την αξιολόγηση. Νομίζω ότι η πρόταση να υπάρχει μια προθεσμία 24 ωρών για την δημοσίευση της αξιολόγησης είναι ευπρόσδεκτη διότι αυτό θα εισαγάγει και το βασικό στοιχείο της διαφάνειας στην όλη διαδικασία και θα διευκρινίσει ότι το περιεχόμενο της αξιολόγησης σχετίζεται άμεσα με τις αντίστοιχες ακροάσεις. Νομίζω ότι ξέρετε εδώ γιατί μιλάω, δεν χρειάζεται να πω κάτι περαιτέρω. Επιπλέον η Επιτροπή θεωρεί ότι το να έχουμε σαφείς και διάφορους κανόνες για ακροάσεις οι οποίες δεν κατέληξαν σε κάποιο συμπέρασμα θα ήταν το ιδανικό. Ε, και πάλι είχαμε ε, τα της διαδικασίας, αυτά αποφασίζονται σε επιτροπές, ορισμένες φορές υπήρχαν κάποιες ακροάσεις οι οποίες θεωρήσαμε ότι δεν κατέληξαν σε σωστά αποτελέσματα. Ε, αν υπήρχαν κάποιες καθορισμένες διαδικασίες θα ήταν πολύ πιο εύκολο εξ αρχής να έχουμε πιο σαφείς διαδικασίες. για την ε, προφορική τροπολογία του κύριου Ντάφ ε, ήδη ανέφερα κάποια πράγματα. Θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξη της Επιτροπής σας για την τροπολογία αυτή, γιατί νομίζω ότι θα ρυθμίσει το θέμα των δυνητικών ε, διαθεσμικών εντάσεων και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο που το, το παρουσίασε ο κύριος Νταφ αφενός σέβεται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους συμπεφωνημένους κανόνες και αφετέρου αυξάνει τη διαφάνεια και την καλύτερη κατανόηση της, όδιας, της όλης διαδικασίας. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν να υποστηρίξετε αυτή την τροπολογία. Θεώρησα ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Τώρα, έχουμε κάποια επιπλέον στοιχεία της έκθεσης. Ο κύριος Νταφ ε, πρότεινε στην αρχική παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ιδέα του Συμβουλίου θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και θα πρέπει να προσκληθεί και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, παρουσίαση αυτή. Ε, και εμεί ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να έρθει όλο το Συμβούλιο όπω είχε προταθεί για να παραστεί σε αυτή την ε, τελετή ε, και φυσικά η πρόσκληση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι απλώς μια ένδειξη ευγένεια από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου τώρα να ολοκληρώσω για το σημείο αυτό και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφ ε, για την έκθεσή του. Όπως θα διαπιστώσετε είναι ελάχιστα τα σημεία διαφωνίας. Σε γενικές ε, γραμμές υπάρχει σύγκληση απόψεων. Συμφωνούμε με τον τρόπο με τον οποίο είδε την όλη διαδικασία ο συγητής και ε, ξέρουμε ότι όλη η διαδικασία είναι απαιτητική και πολύ σημαντική για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επομένως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί τον εισηγητή για τα όσα έκανε και την έκθεση που παρουσίασε. Επιτρέψτε μου τώρα κύριε Πρόεδρε να συνεχίσω με κάποια επιπλέον σχόλια για το διαφθρωμένο διάλογο και την ε, διοργανική συνεργασία. Εδώ επιτρέψτε μου να επισημάνω την ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαίσιο μέχρι τούδε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ε, κατά τη διάρκεια της συζήτηση της συμφωνίας πλαίσιο ε, παρουσιάστηκαν εντάσεις, ε, αμφιβολίες, υπήρχαν και πολύ σοβαρές επιφυλάξεις από πλευρά Συμβουλίου, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ε, ε, τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία πλαίσιο, ήταν γενικότερη ικανοποίηση και παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ ζωηρές οι συζητήσεις στην διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών και αποκλίναμε λίγο από τα προβλήματα τα οποία θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ σημαντικά τότε όταν ε, υιοθετήθηκε η Συμφωνία Πλαίσιο και περάσαμε στα νέα προβλήματα. Είναι σαφές λοιπόν ότι αυτά τα οποία τότε θεωρήσαμε ότι θα ήταν τα πιο περίπλοκα προβλήματα και θα δυσχέρεναν την ε, αμοιβαία συνεργασία μας βρήκαν τη λύση τους και τώρα άκουσα κάποιες επιφυλάξεις στη συνεδρίαση CCC η οποία είχαν σχέση περισσότερο με τις διαβαθμισμένες πληροφορίες ε, και εκεί και η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούν να αναβαθμίσουν την αντιμετώπιση των εγγράφων αυτών σε διεθνή πρότυπα ώστε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση και καλύτερο χειρισμό των διαβαθμισμένων αυτών εγγράφων, κάτι που είναι προ όφελο και των δύο οργάνων και νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο πολύ σύντομα, διότι η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπή και Κοινοβουλίου επί του θέματο ε, είναι πολύ καλή. Δεύτερον θέμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικώς τον ε, πρόεδρο Καζίνη, συνεργασία για το Μητρό Διαφάνειας, όπου και πάλι η πραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, διότι μας έδωσε καλές απαντήσεις, καλές λύσεις ε, στα πολύ περίπλοκα ζητήματα του πώς μπορούμε να μετατρέψουμε κάτι το οποίο είχε θεωρηθεί ως ε, Μητρό Ομάδων Συμφερόντων ε, σε εργαλείο ε, υπέρ της διαφάνειας στις Βρυξέλλες. Πώς μπορούμε να το διαβρύνουμε ώστε να συμπεριλάβουμε και άλλες πτυχές του πολιτικού χώρου στις Βρυξέλλες που δεν είναι λομπίστες αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να είναι δραστήριοι στην πολιτική συζήτηση στις Βρυξέλλες και χάρη στην καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τη διαπραγματευτική ομάδα νομίζω ότι το επιτύχαμε αυτό και το μητρό διαφάνειας θα είναι αυτό το οποίο θα ε, κάνει την αλλαγή για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις ομάδες συμφερόντων στις Βρυξέλλες και πώς όλοι οι φορείς που προσπαθούν να είναι δραστήριοι στην πολιτική συζήτηση σε ευρωπαϊκά θέματα θα είναι γεγραμμένοι ε, με διάφανο και θετικό τρόπο. Γνωρίζω ότι τώρα θα αρχίσει η συνεργασία για το πώς ε, θα μπορέσει να συμμετέχει το Συμβούλιο στο Μητρό. Είμαι αισιόδοξο ότι θα επιτευχθεί ο στόχο αυτός και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα το γεγονός ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα μπορούν να συμφωνήσουν επί του θέματος και θα ε, υπερτονίσουν τη σημασία της διαφάνειας ε, στον τομέα αυτό του Μητρό Διαφάνειας. Τέλος. Έγιναν πολύ έντονε συζητήσει στη διάρκεια τη προηγούμενη Ολομέλεια για την τροποποίηση της συνθήκης και τον τρόπο με τον οποίο θα έχουμε αυτό το νέο στοιχείο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και εδώ με τα χαράς μπορώ να σας δηλώσω ότι παρά τις απαιτητικέ ε, θέσεις και τις ε, αυστηρές αρχικές θέσεις κάποιων κρατών μελών εξ αρχής, τώρα μετά από τη Σύνοδο της Ευρωζώνης την Παρασκευή κατέστη σαφές ότι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη συνοχή μεταξύ του μηχανισμού σταθερότητας και την οικονομική διακυβέρνηση και θα μπορέσουμε να έχουμε όλε τι ευρωπαϊκέ αρμοδιότητε και να διασφαλίσουμε τον κεντρικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλο το νέο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα το οποίο θα πρέπει να δομήσουμε για την οικονομική διακυβέρνηση και τη στενότερη οικονομική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά για την προάσπιση του κοινού μα νομίσματο. Νομίζω ότι επετέφθη ο στόχο και ε, η αρχική θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Κοινοβουλίου και η στάση που τήρησαν σε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση ήταν η ορθή και καταφέραμε να διαμορφώσουμε τη συζήτηση κατά τρόπον ώστε να σέβεται πολύ σαφώς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συνεργαζόμαστε σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και σε αυτό το τόσο σημαντικό τομέα στο μέλλον. Τελευταία σχόλια για τον ε, διαρθρωμένο διάλογο. Χαίρομαι για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο διάλογος με τους επιτρόπους και τις αρμόδιες επιτροπές. Προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε αυτό το νέο στοιχείο στο πρόγραμμα εργασίας τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στα επόμενα χρόνια, αλλά σας ενημερώνουμε και εσά και το ευρύ κοινό. Τι προγραμματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέσα επόμενα χρόνια. Περίπου εκεί κοντά στο τέλος της ε, θητείας της. Βλέπετε ότι είναι συγκεκριμένη κουβέντα, οπότε και έχουμε προβλεψιμότητα του προς τα που θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και γι' αυτό και μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν τον ε, διαρθρωμένο διάλογο και με τους, Ευρωπαϊκούς, και με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους και επομένως την Άνοιξη θα έχουμε τη συνάντηση με τους Πρόεδρους των Επιτροπών και θα έχουμε και το σχετικό ψήφισμα εκείνο το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το ζήτημα, γιατί όλα αυτά είναι συστατικά πολύ σημαντικά για το δικό μας ε, πρόγραμμα εργασιών του 2012. Ακριβώς όπως ε, ε, πρόκειται να ενεργηθούν τα πιο συγκεκριμένα κομμάτια της διαδρομής το Σεπτέμβριο φέτος. Έτσι επομένως σιγά σιγά υλοποιούμε το πρόγραμμα των ενεργειών μας εν ώψη της στρατικής του 2020 και θα και την πρώτη χρονιά που πιστεύουμε θα χρησιμοποιήσουμε τα νέα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και έτσι θα έχουμε την καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση, καλύτερη προσπάθεια συντονισμού και έτσι θα προσανατολίσουμε και τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις οικονομικές τους επιδόσεις. Βεβαίως έχουμε και του στόχους μας του προγράμματος της Στοκχόλμης ούτως ώστε να ενισχύσουμε την έννοια αγορά. Ξέρω ότι πιέζει ο χρόνο, ότι είναι πολύτιμο για την επιτροπή σα. Εδώ θα βάλω τελεία και ευχαρίστω να απαντήσω τυχόν ερωτήσει. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε ο Έχει δει το λόγο κύριο Γκερέρο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε επίσης. Ξέρετε, έχω διατελέσει σκιώδης για την έκθεση DAF. Είμαι σκιώδης και όλοι συνεργαζόμαστε με τον κύριο DAF και είμαστε πάρα πολύ συντονισμένοι έχει δημορφωθεί ευρεία συνένεση για το ε, δουλειά μας. Πάντως, πέραν αυτών, εγώ έχω διατυπώσει κάποιες συγκεκριμένες ε, τροποποιήσεις τη εκθέσεις DAF. Αυτές τις τροπολογίες θέλω να προτείνω ε, κάποιες ιδέες μου για τα θέματα που και εσείς αναφέρετε κύριε Επίτροπε και είπα ότι ούτε για 20 ούτε για 10 λεπτά είπα για 15 λεπτά. Δηλαδή για να βρεθεί η μέση οδός. Και επομένως ο υποψήφιος επίτροπος να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να έχει κάποιο χρόνο αρκετό αλλά και από την άλλη μεριά να μην τρώει πάρα πολύ χρόνο. από την ε, ακρόαση. Ε, η άλλη μου πρόταση αφορούσε το ότι μέσα σε αυτό το τρίωρο να δούμε τι θα γίνει αν δεν καταλήξουμε σε συμπέρασμα, συμπέρασμα ξεκάθαρα ή αν θα μπορούσαμε να έχουμε, να, θέλουμε, να θέλουμε και άλλες πληροφορίες από τον υποψήφιο ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα να συγκληθεί μια νέα συνάντηση της Επιτροπής και να μπορούμε να εξετάσουμε και άλλο τον υποψήφιο. Κάτι άλλο τώρα το οποίο μου ήλικε την προσοχή είναι ο αναβαθμιμένος ρόλος των συντονιστών όλων των πολιτικών πτέρυγων του Κοινοβουλίου για την οργάνωση αυτών των ε, ακροάσεων. Βεβαίως και ο κάθε βουλευτής εξετάζει όπως νομίζει τον υποψήφιο, αλλά η εμπειρία μου λέει ότι συχνά διατυπώνουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Και ο βουλευτής που είχε κατά νου να υποβάλει μια ερώτηση, την υποβάλλει κι ας ήδη την έχουν υποβάλει την διαρώτηση άλλοι τρεις προηγουμένως. Άρα θα μπορούσε να γίνει μια συνάντηση συντονιστών και να υπάρξει ανταλλαγή των ε, ερωτήσεων του τι ενδιαφέρει κάθε πολιτική ομάδα. Και έτσι να γίνει μια κατανομή της δουλειάς. Και αντίστοιχα κατανομή των ερωτήσεων αναβουλευτή και αν ακόμα Και καθένας να διαλέξει πού θέλει διευκρινήσεις, πού θέλει απαντήσεις από τον υποψήφιο. Τέλος. Άλλη δυνατότητα θα μπορούσε να είναι για, για την κατάληξη της ακρόασης, για την επιστολή αυτή, να υπήρχε κάποιο συζητητή στην ε, αντίστοιχη επιτροπή και αυτός ο εισηγητής να έχει έτσι εξέχοντα ρόλο, κατοχυρωμένο, θεσμικό α το πούμε έτσι, στις ακροάσεις. Ναι, με συμφωνείτε και εσείς για την θεσμική οποία που να πετύχουμε και οπότε θα πρέπει να δούμε και εγώ θα μπορούσα να σας διευκρινίσω ότι θέλετε. Όμως αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι το ότι υπάρχει τελικά και κάποια ενδιάμεση κατάσταση κατά την οποία δεν καλείται ο υποψήφιος πρόεδρος να εξηγήσει πώς ε, κατένει με τα χαρτοφυλάκια στους υποψηφίους. Αλλά να μπορεί να προσκληθεί αυτός ο πρόεδρος της Κομισιόν και να εξηγήσει τα γενικότερα κριτήρια για την συγκρότηση του Σώματος Επιτροπής σε σχέση με το πρόγραμμα το οποίο έχει παρουσιαστεί στην Ελλομέλεια και σε σχέση και με τις ε, προτεραιότητες. Έτσι ο ρόλος, η προσέλευση του Προέδρου της Επιτροπής δεν θα συνιστούσε έλεγχο όσον αφορά την κατανομή των χαρτοφυλακίων. Θα ήταν ένας διάλογος, μια συζήτηση. Απλώς θα γινόταν μια ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τα γενικότερα κριτήρια. Σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες, επομένως, που έχει τάξει ο Πρόεδρος ε, όταν μίλησε στο Κοινοβούλιο. Τώρα, για το δεύτερο τμήμα που μας είπατε, να εξαντλήσουμε όλα όσα προσφέρει η συνθήκη. Σύμφωνα με και τόσα είπαν στην ένταση κορυφή την προηγούμενη εβδομάδα. Και έτσι η Ολομέλεια να δώσει το πράσινο φως για την αποσταθμένη μορφή της συνθήκης. Όταν εξασφαλιστεί ο έλεγχος, ε, η λειτουργία αυτού του μηχανισμού σταθερότητας. και όχι μόνο ως προς τις χώρες της Ευρωζώνης, αλλά και όσον αφορά την κατοχήρωση του συντονιστικού ρόλου Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Yes, thank you very much. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε και μας δώσατε αυτή την γενική εικόνα για τις ακροάσεις. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, νομίζω όλοι είμαστε ικανοποιημένοι με την έκθεση του Ανδρίου Νταφ, η οποία είναι ευρύτατη και εις βάθος και κάνει καλές συστάσεις. Νομίζω πως ε, επίσης ε, λογικό είναι να μην ε, συζητάμε μόνο με τους ε, ορισμένους επιτρόπους αλλά να ξεκινήσουμε μια ανταλλαγή απόψεων και με τον ε, ορισμένο πρόεδρο της Κομισιόν για τις γενικές ιδέες στελέχωσης της Κομισιόν και θεωρώ επίσης πως υπάρχει μια υποχρέωση από πλευρά των ορισμένων επιτρόπων να προετοιμαστούν, αλλά υπάρχει και υποχρέωση δική μας να προετοιμαστούμε στο δυνατόν καλύτερα για να μην γίνεται δύο φορές ή τρεις και τέσσερις και πέντε η ίδια ερώτηση. Και συμφωνώ με την ιδέα πως θα πρέπει να υπάρχει μια προπαρασκευαστική ε, ομάδα συντονιστών για να είμαστε προετοιμασμένοι και να υπάρχει μια συνέχεια στην ακρόαση. Μπράβο με τις ευκαιρίες ε, για να σας ρωτήσω τι έχει γίνει για την θέση ενισχύ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και από πλευράς της Κομισιόν και όσον αφορά το προσωπικό που χρειάζεται για τις τεχνικές, νομικές και πολιτικές πτυχές της ε, διαδικασίας και βεβαίως όσον αφορά την διαδικασία προετοιμασίας της κύρωσης ε, στα κράτη-μέλη, ειδικά όταν μιλάμε για τα ζητήματα της επαλήθευσης και ειδικά εάν δούμε ακόμα, τις προβληματικές ακόμα πτυχές της διαδικασίας online που υπάρχουν στον κανονισμό. Αυτό είναι το σημαντικότερο για την ώρα. Τελευταία ερώτηση σύντομα. Να σας ρωτήσω. Τι άποψη έχετε για τα θεσμικά και τα συνταγματικά και τα διοικητικά της Κομισιόν. Τι άποψη έχετε για την πρόταση αυτή για το μηχανισμό σταθερότητας, πώς θα πρέπει τώρα να λειτουργήσει, να συσταθεί, γιατί φοβόμαστε πως έχει συσταθεί εκτός της κοινοτικής μεθόδου και των θεσμικών οργάνων, ειδικά της Κομισιόν που έχει γνώση και ικανότητα να δει τα ζητήματα αυτά. Οπότε αν θα θέλατε να σχολιάσετε, ευχαριστώ να σας ακούσω. Ο κύριος Νταφ ζητάει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όσους μίλησαν ε, για την έκθεση. Ε, Κύριοι Γκερέρο και Σεύσοβιτς έχουν δίκιο όταν λένε πως τα 15 λεπτά είναι πιο κατάλληλος χρόνος για την αρχική δήλωση ε, ενός εκλεγμένου επιτρόπου από τα 10 που έχω εγώ. Συμφωνώ με τον Επίτροπο πως κάθε εκλεγμένος Επίτροπος πρέπει να έχει ίδια μεταχείριση και άρα ίδιο χρόνο ακρόασης. Συμφωνώ πως η ευθύνη των συντονιστών πρέπει να ενισχυθεί ή δυνατόν. Αν και σε τελική ανάλυση ε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τους ευρωβουλευτές που δεν έχουν πειθαρχία, εξάλλου εδώ μέσα είναι κοινοβούλιο. Όχι κανένα τάγμα πεζικού. Οπότε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα βελτιώσουμε την όλη διαδικασία. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σεφτσεβίτς για τον κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί όπως ξέρει αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για την διαδικασία έγκρισης της Κομισιόν. Στο σχέδιο στην παραγραφό 1.5 μιλάει για τη δήλωση συμφερόντων και λέει πως η δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται όταν το μέλος της Επιτροπής αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Αυτό είναι αργά. Χρειάζεται δήλωση αυτή συμφερόντων πριν την αρχή των ακροάσεων και προτείνω να τις, εξετάσει, να τις εξετάζει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σε ένα πρώτο βαθμό και μόνο σε περίπτωση αμφιβολίας ή ασυνεπιών ή κάτι, κάποιες τέτοιες περίπτωσης μόνο σε αυτή την περίπτωση οι τομεακές επιτροπές που είναι υπεύθυνε για την ακρόαση θα θίγουν το ζήτημα της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. Είναι σημαντικό να υπάρχει μία ενιαία προσέγγιση εναντί όλων των επιτρόπων όσον αφορά τη δήλωση. και εγώ ζήτησα η διάσκεψη των Προέδρων να θέσει αυτό το θέμα όταν θα συζητήσουν τον κώδικα συμπεριφοράς με τον Πρόεδρο Μπαρόζο και θα ήθελα να γνωρίζω το αποτέλεσμα του ετήματος αυτού για να δω αν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την παράγραφο. Για να επιμείνουμε στο ότι θα πρέπει να συμπληρώνει τη δήλωση η Επιτροπή πριν την ακρόση. Για το θέμα του μηχανισμού σταθερότητας, όπως ξέρετε, η Επιτροπή μας, παρά το ότι δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα στην Ολομέλεια, πρότεινε οι κανόνες για τη λειτουργία του μηχανισμού να συνταχθούν σε έναν κανονισμό δηλαδή να τους προτείνει η Κομισιόν και συναπόφαση να αποφασίσει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και Νομίζω πως οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να συμπεριλάβουν αυστηρούς όρους που, αυτούς που αναφέρονται στο σχέδιο αλλαγής ε, της συνθήκης και θα ήθελα να επιβεβαιώσουμε πως ο πρόεδρος Μπαρόζο στις ε, συναντήσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα στηρίξει το Κοινοβούλιο στο συγκεκριμένο αίτημα κανονισμού για να λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός παρά το ότι ο μηχανισμός ο ίδιος ε, θα ε, συσταθεί με διακυβερνητική συνθήκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για την απάντηση θα λάβει τον λόγο ο κύριο Σεύκολτς, αλλά θέλω και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η πρώτη μου παρατήρηση αφορά τα πολιτικά κόμματα. Σήμερα το πρωί Ψηφίσαμε την έκθεση της κυρίας Γεννάκου για την εφαρμογή του κανονισμού 2004-2003 για την ε, χρηματοδότηση και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την Επιτροπή μας και θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να κάνει και προτάσεις επί του θέματος. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση της οποίας ο εκλογικός νόμος ε, είναι μια πολύ σημαντική πτυχή, χρειάζεται και ευρωπαϊκά κόμματα, κόμματα συγγνώμη, τα οποία θα είναι πραγματικά ευρωπαϊκά. Αυτή είναι η πρώτη με ερώτηση. Το δεύτερο αφορά το διαρθρωμένο διάλογο. Όπως σας είπα προηγουμένως, εμείς ως Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων δεν έχουμε μεγάλες ε, νομοθετικές αρμοδιότητες. Έχουμε όμως συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε θέματα διοργανικών συμφωνιών. Και το άρθρο 17 σημείο 1, τελευταία παράγραφος, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά τη ε, διαδικασία του ετήσιου προγραμματισμού για να καταλήξει σε διοργανικές συμφωνίες. Όχι τόσο ως προς την ουσία, αλλά ως προς τη μέθοδο, η Επιτροπή μας είναι ε, η αυτή η οποία έχει καθήκον να παρέμβει. Ευχαριστώ και σας ζητώ το λόγο τώρα. Σας δίνω το λόγο τώρα, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές, τα μέλη της Επιτροπής που μίλησαν. Ξεκινώντας με τον κύριο Γκερέρο. 15 λεπτά νομίζω είναι ένας λογικός συμβιβασμός γιατί εάν κάθεται κανείς ε, και υφίσταται μία ακρόαση, τα πρώτα δέκα λεπτά περνάνε γρήγορα στην παρουσίαση και μετά βεβαίως τα επόμενα πέντε λεπτά να απαντά ερωτήσει δεν περνάει η ώρα. Οπότε 15 λεπτά νομίζω είναι λογικός χρόνος και Νομίζω πως ε, και οι συνάδελφοι του Επιτροπή πέρασαν κάτι παρόμοιο και οπωσδήποτε μελλοντική επιτροπή θα εκτιμήσουν τις προτάσεις αυτές. Συμφωνώ επίσης με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γκερέρο και ο κύριος Χέφνερ για την προετοιμασία και των δύο πλευρών. Πράγματι, οι ορισμένοι, οι διορισμένοι επιτροποί πρέπει να έρχονται προετοιμασμένοι και πρέπει εδώ πέρα να δείξουν πως είναι ικανοί για το αξίωμα αυτό πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία αποτελούν τμήμα των χαρτοφυλακίων, πώς θα είναι καλή πολιτική εταίροι των επιτροπών. Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούν το δυνατόν περισσότερο σε σύντομη ε, συχνά χρονική περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ ορισμού και ακρόασης και καλό θα είναι μια αναλογική προετοιμασία να γίνεται και από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αποφύγουμε ε, τις ίδιες ερωτήσεις ή να προσπαθήσουμε λίγο πολύ να συζητήσουμε με τους συντονιστές για το πώς θα δομηθούν οι ερωτήσεις ειδικά αν είναι ευρύτερο το χαρτοφυλάκιο και έχει πολλούς τομείς ευθύνης για να είναι έτσι και όπως πιο συνεκτική συζήτηση. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο είπε ο Άντριου Ντάφ, ότι εδώ πέρα είναι κοινοβούλιο και ο οποιοδήποτε, οποιοδήποτε βουλευτής μπορεί να ρωτήσει οτιδήποτε. Αλλά αν υπάρχει καλύτερη προετοιμασία, οργάνωση, νομίζω θα είναι πιο καλό για την ακρόαση και για τους ευρωβουλευτές και για το κοινό και νομίζω πως θα επιτρέψει στον Επίτροπο να παρουσιάσει μια πιο πλήρη εικόνα για το τι θα ήθελε να κάνει στον τομέα αυτόν γιατί θα μπορέσει να μιλήσει για τον ίδιο τομέα απαντώντας πολλές ερωτήσεις. Οπότε νομίζω πως θα είναι αμοιβαία υποφελές η ιδέα τώρα ε, περί ενός εισηγητού της ακρόασης θα είναι θετικό γιατί θα φροντίζει τη διαδικασία με μεγάλη λεπτομέρεια και θεωρώ επίσης πως η διαδικασία της εξπόστα αξιολόγησης ε, νομίζω ολοκληρώθηκε και ε, θα ολοκληρωθεί έτσι καλύτερα όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Γκερέρο νομίζω πως είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει κάποιες ερωτήσεις στον πρόεδρο, στον εκλεγμένο πρόεδρο της Κομισιόν για τη φιλοσοφία του, για το ποια θα είναι τα γενικά κριτήρια, για τις απόψεις του ή της, ε, για την κατανομή μελλοντικών ε, χαρτοφυλακίων ε, σε μια ολομέλεια. Νομίζω καλό είναι να γίνουν όλα αυτά εκ των προτέρων ε, έτσι ώστε να μπορεί να παρουσιάσει την φιλοσοφία του, την προσέγγιση του ο εκλεγμένος πρόεδρος ήδη σε εκείνη τη χρονική στιγμή και καλό θα είναι και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξέρει τι φιλοσοφία ε, έχει στην στην κατανομή των χαρτοφυλακίων ο πρόεδρος της ε, Κομισιόν. Τώρα γιατί μου άρεσε η προφορική τροπολογία DAF γιατί σέβεται την ε, συνθήκη, τη διοργανική ισορροπία και ε, βεβαίως παραμένει το προνόμιο της κατανομής των χαρτοφυλακίων από πλευράς Πρόεδρου της Κομισιόν. Οπότε δεν δημιουργείται εδώ πέρα η δυνατότητα διαπραγμάτευσης για το ποιος ε, θα λάβει τι. Οπότε, ξέρετε, ξέρετε τι λέω. Θα φτάσουμε σε μια διαδικασία που μετά θα ήταν μεγάλο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Γιατί νομίζω πως είναι δικαίωμα του εκλεγμένου Προέδρου να αποφασίσει πως ε, θα διανύμει τα χαρτοφυλάκια και ποιοι είναι οι καλύτεροι υποψήφοι και μετά βέβαια θα πρέπει να έρθει ενώπιόν σας και να αποδείξει πως είναι ικανή για αυτές τις δουλειές και αντάξει της εμπιστοσύνη σας γιατί νομίζω έτσι είχε σχεδιαστεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και έτσι μοιράζονται οι ρόλοι. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Γκερέρο για τα σχόλιά σας για την αλλαγή της ε, συνθήκης και την απλοποιημένη διαδικασία. Όπως σωστά επισημάνατε είναι πολύ σημαντικό στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα θα δημιουργήσει επιπλέον μέσα για την οικονομική σταθερότητα, την υπεράσπιση του ευρώ και τη δημιουργία αυτού το οποίο θα θεωρούσα σε κάποια κράτη-μέλη ως πλήρη νομική βεβαιότητα και πως όλα αυτά θα συμμορφώνονται πλήρως και με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις εθνικές συνταγματικές τάξεις είναι κάτι το πολύ σημαντικό και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα γιατί αν ακολουθήσουμε την τακτική ε, διαδικασία θα βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη συζήτηση που θα αφορά πιθανές ε, ε, μεταφορές αρμοδιοτήτων ε, φυστάμενες ή ε, στην αντίληψη των ανθρώπων μόνο και μετά θα περιπλακούν πολύ τα πράγματα οπότε έτσι πρέπει να κινηθούμε και ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ότι είναι διατεθειμένο να στηρίξει την προσέγγιση αυτή. Ε, απαντήσω τώρα στον κύριο Χέφνερ ειδικά στο δεύτερο και τρίτο κομμάτι των ερωτήσεων όσον αφορά την Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία Πολιτών στην οποία συνεργαστήκαμε. Εγώ χαίρομαι για το ότι αν μιλήσουμε για αυτά τα οποία θα κάνει η Κομισιόν, ειδικά τη δημιουργία του site και την προετοιμασία του ανοιχτού λογισμικού, του λογισμικού ανοιχτού κώδικα που θα επιτρέψει στους οργανωτές να κατεβάσουν το λογισμικό δωρεάν και να το χρησιμοποιήσουν για τη συλλογή υπογραφών που θα στηρίζουν τις πρωτοβουλίες αυτές ε, δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως θα τα καταφέρουμε και τα δύο εγκαίρως ε, και έχουμε προχωρήσει αρκετά και δεν νομίζω πως θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουν λυθεί τα προβλήματα του software ε, πριν τεθεί ενισχύει ο κανονισμός ε, το επόμενο έτος και το ίδιο μπορώ να πω βεβαίως και για το εγχειρίδιο το οποίο θα έχει προετοιμαστεί για το ότι όταν θα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν οι οργανωτές ήδη από την 1η Απριλίου 2012 θα έχουν όλες τις πληροφορίες εκ των προτέρων και θα μπορούν να προετοιμαστούν αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο μέσο δημοκρατικού διαλόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την κατάσταση στα κράτη-μέλη μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Νιώθουν την ίδια δημοκρατική πίεση που νιώθουμε και εμείς στην Κομισιόν. Ναι. και για το καλό τη κοινωνία των πολιτών θα τεθεί ενισχύ εγκαίρω το μέσο αυτό και όλες οι νομικέ αλλαγέ στο εθνικό επίπεδο θα γίνουν. Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, θεωρώ πως ε, συμφωνούμε εδώ πέρα. Εμείς θεωρούμε πως θα μπορέσουμε να βρούμε λύση στο πλαίσιο των συνθήκων Επίσης ε, θα προετοιμάσουμε το να έχουμε τον Εθνικό Μηχανισμό σταθερότητα στο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαχείριση αυτής της πολύ σημαντικής διαδικασίας και να είναι αποδεκτό από τα κράτη-μέλη. Οπότε, όπως πολλές φορές ε, έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να αναζητήσουμε έναν ε, συμβιβασμό και νομίζω πως ε, τελικά καταφέραμε να έχουμε ένα συμβασμό αποδεκτό γιατί εκπληρώνει τον ρόλο του μηχανισμού ε, σταθερότητας και βέβαια πρέπει να γίνει σύμφωνα με την συνθήκη και σε διαφορετικά επίπεδα, είτε μιλάμε στο Συμβούλιο, είτε στον Πρόεδρο τη Κομισιόν και να γίνει και όλη η προπαρασκευαστική τεχνική εργασία. Η Κομισιόν δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει το προνόμιο της αν θεωρούν πω ξεφεύγουμε από το πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου γιατί είναι κάτι το σημαντικό, αναγκαίο και ε, βεβαίω ε, θα πρέπει να σεβόμαστε τις συνθήκες και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν την εξέλιξη της διαδικασίας. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το ρόλο μας. Να υπάρχει συνοχή στην ευρωπαϊκή πολιτική και να παίξουμε τον κεντρικό ρόλο που μόνο η Κομισιόν μπορεί να παίξει για αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τομείς όπως η οικονομία, η ανταγωνιστικότητα, η δημιουργία πολιτικών για νέες σύγχρονες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Ντάφα για τον κώδικα συμπεριφοράς, η συζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων ήταν επικοδομητική και συγκεκριμένα όταν μιλάμε για την δήλωση των συμφερόντων αυτό το οποίο προτείναμε είναι πως πρέπει να υπάρχει ανανέωση κάθε χρόνο και βεβαίω να αφορά και τον την σύζυγο ή σύντροφο. Οπότε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων βεβαίως θα πρέπει να έχει πριν από την ακρόαση τη δήλωση. Εγκλαμβάνουμε αυτό το οποίο λέτε πράγματι. Αναμένουμε τώρα την ε, γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα υιοθετηθεί από διάσκεψη των Προέδρων. Φαντάζομαι πως αυτό θα περιέχεται στην γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως ε, θα το φέρω αυτό στο σώμα των επιτρόπων γιατί πράγματι αντιλαμβάνουμε γιατί πρέπει να υπάρξει αυτή η αλλαγή όσον αφορά το πώς ε, θα διαχειριστούμε το μηχανισμό σταθερότητας και το πώς θα έχουν οι εσωτερικές διαδικασίες Βλέπω τις προτάσεις σας εδώ πέρα για κανονισμό, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δεσμευτώ για κάτι, γιατί δεν μπλέκομαι εγώ στο χαρτοφυλάκιο αυτό. Πρέπει να συσκεφθώ με τους συναδέλφους, να δούμε... <coughs> θα γίνουν αυτές τις προτάσεις και πώς θα γίνουν αποδεκτές. Έχουμε ένα γενικό σχέδιο αυτή τη στιγμή για το πώς θα έχουμε και την ευθύνη των ιδιωτών, επενδυτών, ποιες ε, συλλογικές ρήτρε ε, μπορούν να εισαχθούν στο μηχανισμό και ποια θα είναι αυτή η λεπτή γραμμή μεταξύ ελεγγύης και αποφυγής του ηθικού κινδύνου και βεβαίως συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Και ξέρετε πως ε, όλοι αυτοί οι νέοι κανόνες που αναμένουμε είναι στο παράρτημα 2 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου και νομίζω πως η συζήτηση δεν έχει ακόμα φτάσει στο πως θα είναι οι εσωτερικές διαδικασίες του μηχανισμού όσον αφορά την τελευταία παρέμβαση του κυρίου Κασίνη στα πολιτικά κόμματα Αναμένουμε βεβαίως ακόμα την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μπορώ να πω πως έχουμε ένα κοινό στόχο. Αυτός είναι η φελτίωση, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού δημοσίου χώρου. Οπότε, αν θεωρείτε πως οι κανονισμοί του 2003 και 2004 χρειάζονται ανανέωση, ε, ευχαρίστω να το συζητήσουμε αν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Ε, έρθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Τέλος, προγραμματισμός της Ένωσης. Αυτό το συζητήσαμε και στη Συμφωνία Πλαίσιο. Θεωρώ πως ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε με τον προγραμματισμό είναι πολύ συγκεκριμένες συζητήσεις των τριών ε, θεσμικών οργάνων Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιών για το πώς θα δοθεί προτεραιότητα στο έργο μας για την επόμενη ε, περίοδο γιατί αυτός θα είναι ο καλύτερος συμβιβασμός μεταξύ του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας της Κομισιόν αφενός και αφετέρου της εμπλοκής του νομοθέτη για τα κυριότερα ζητήματα προτεραιότητα του επόμενου έτους γιατί έτσι θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε καλύτερα τον χρόνο των συζητήσεων της έγκρισης, καλύτερο συντονισμό του έργου του νομοθέτη και των δύο νομοθετικών σωμάτων και θα έχουμε έτσι καλύτερα αποτελέσματα εκεί όπου τα χρειαζόμαστε. Για να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα λοιπόν για τι προτεραιότητε της Ένωσης αυτό το έτο είναι το πακέτο οικονομικής διακυβέρνηση και εύκολα θα συμφωνήσουμε σε αυτό και έτσι νομίζω είναι, αυτό είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία και θα καταλήξουμε νομίζω σε παρόμοια συμπεράσματα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ελπίζω φέτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε, το γεγονός ότι είστε πάντα ευπρόσδεκτος εδώ. Νομίζω ότι με τις τελευταίες ευχές μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς έχουμε ένα ακόμα θέμα να συζητήσουμε. Αν θέλετε να φύγετε μπορείτε κάλλιστα να φύγετε. Αν θέλετε να μείνετε με τα χαράς. Εμείς έχουμε ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη, αλλά νομίζω ότι λείπει ο νομικός θα σας κάνω μια παρουσίαση του σημείου, θα σας προτείνω την ε, ε, άκουσα που θέλουμε να ακολουθήσουμε, που θέλουμε να αποστείλουμε μία επιστολή για το άρθρο 128 και επειδή δεν έχουμε παρκεριθμό μελών, να δούμε ποιος θα ψηφίσει. Ο κύριος ε, Λάινεν έχει ζητήσει να δούμε κατά πόσον μπορούμε ε, να έχουμε μία εξέταση του θέματος. Έχουμε το άρθρο 228 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν διαβάσουμε μαζί το σημείο αυτό, εντάξει είναι λίγο ανιαρό το να διαβάζει κανείς το, τα άρθρα του κανονισμού, αλλά ίσως θα έπρεπε να διαβάσουμε μαζί τις διατάξεις για να δούμε και την ερμηνεία τους. Το άρθρο 128 λοιπόν του κανονισμού μας αναφέρεται στις προσφυγές στο ε, δικαστήριο, δηλαδή προσφυγές του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το άρθρο 128 λέει, υπαριθμόν 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός των ε, ορίων που καθορίζονται από τη συνθήκη και του καθεστώτος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τι προσφυγές των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωση ή φυσικών ή νομικών προσώπων εξετάζει την ομοθεσία τη Ένωση και τα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συνθήκε κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου, γίνονται απολύτως σεβαστά. Εδώ λοιπόν η δυνατότητα προσφυγής ε, γίνεται υποδεικνύοντας την νομοθεσία και τις διαδικασίες δράσης. Το άρθρο 228, σημείο 11, Ναι, ναι, το 11 είναι. Τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι ένα κράτο μέλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να ζητήσουν τη γνωμοδότηση του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ε, ταύτιση μιας προβλεπόμενης συμφωνίας με τις συνθήκες. Εάν το δικαστήριο δώσει αντίθετη γνώμη, τότε δεν μπορεί να ισχύσει η συμφωνία. Η συνθήκη λοιπόν αναφέρεται στη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμάς μας ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο, να ζητήσουν τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όταν μιλάμε για συμφωνία η οποία προβλέπεται από τις συνθήκες. Συμφωνία. Αλλά δεν μιλάμε για έλεγχο της νομοθεσίας ή έλεγχο των εκτελεστικών πράξεων. Η απάντηση κατ' εμέ είναι πολύ απλή. Καταρχάς θα πρέπει να διαβάσουμε και το άρθρο 90 του κανονισμού, το οποίο άρθρο 90 στο σημείο 7 λέει πριν από την ψηφοφορία για την έγκριση, η αρμόδια επί της επιτροπή και εδώ αναφερόμαστε στις διεθνείς συμφωνίες, έτσι. Πριν από την ψηφοφορία λοιπόν τη αρμόδια επιτροπή, μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 1 δέκατο των Ευρωβουλευτών μπορεί να προτείνουν το Κοινοβούλιο να ζητήσει την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το κατά πόσον είναι συμβατή μια διεθνή συμφωνία με τι συνθήκε. Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση, η ψηφοφορία ε, αναστέλλεται μέχρι την ε, έκδοση της γνωμοδότησης του Κοινοβουλίου. Συγκρίνοντα αυτού του τρει κανόνε, κατά την άποψή μου απορρέουν τα εξή. Πρώτον, ότι η συνθήκη, που είναι ο πρωτογενή κανόνα, ο πρωτογενή νόμο, μα δίνει τη δυνατότητα προσφυγή για τι διεθνεί συμφωνίε. Επομένω, ο κανόνα που εφαρμόζεται εδώ είναι το άρθρο 90 και όχι το άρθρο 128. Με άλλα λόγια, το άρθρο 128 δεν αναφέρεται στις συμφωνίες, αλλά αυτό δεν μας ανησυχεί, γιατί σε αυτό αναφέρεται το άρθρο 90. Πρόκειται για ένα θέμα δηλαδή το οποίο ε, αναφέρεται σε άλλο σημείο του κανονισμού. Το άρθρο 128 αναφέρεται μόνο σε προσφυγή στο δικαστήριο όσον αφορά την νομοθεσία και τις εκτελεστικές πράξεις και δεν αναφέρεται σε άλλες δυνατότητες, ε, θεωρητικές δυνατότητες προσφυγής που είναι οι εκτελεστικές πράξεις και κάποιες άλλες αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν νομοθετική αξία αλλά μπορούν στη θεωρία να παραβιάζουν τις συνθήκες και θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο. Ποιες είναι οι συνέπειες τώρα. Καταρχάς είναι προφανές ότι καθήκον της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου είναι να είναι θεματοφύλακες και να φροντίζουν ότι ε, τα όσα ε, συμφωνούνται είναι σύμφωνα με τη ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση αυτής της αρχής θα πρέπει να μεταγραφεί στον κανονισμό μας. Ο κανονισμός μας όμως δεν μπορεί αντίθετα με αυτή την αρχή να μην δίνει τη δυνατότητα προσφυγή. Επειδή δηλαδή δεν αναφέρεται κάτι στον κανονισμό, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγή. Όσον αφορά τι διεθνεί συμφωνίε, υπάρχει το άρθρο 90 και όσον αφορά τι ε, εκτελεστικέ πράξει και τι άλλε δυνατότητε ε, γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ερμηνεία μα το άρθρο 128 και το άρθρο 128 καθορίζει ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του δικαστηρίου για θέματα νομοθεσίας και εκτελεκτιστικές πράξεις. Μας φαίνεται λοιπόν παράλογο να ε, αποκλείονται η καταξουσιοδότηση πράξης και οι υπόλοιπε νομοθετικές διαδικασίες. Ακολουθώντας λοιπόν τη λογική, στα λατινικά τουλάχιστον, στα, ευρωπαϊκά, στα ε, πανεπιστημιακά εγχειρίδια λέγεται ότι ubi adem registris, ubi adem που σημαίνει ότι θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να μας λέει κατά πόσον μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκό δίκαιο και να ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Επειδή λοιπόν το άρθρο 90 αναφέρεται στο 1 και το άρθρο 128 αναφέρεται στις υπόλοιπες περιπτώσεις, επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αναλογικά βάσει της λογικής ισχύουν και η κατεξουσιοδότηση πράξης και οι υπόλοιπες νομοθετικές πράξεις. Αυτή είναι η λογική του κανόνα και νομίζω ότι πολύ εύκολο θα μπορούσαμε να το παρατείνουμε και να πούμε ότι λογικά αυτό προκύπτει. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω το εξή. Και σα το διαβάζω εδώ, αλλά δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε εδώ γιατί δεν έχουμε απαρτία. Να λάβω την έγκριση να ε, αποστείλω την επιστολή, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η ερμηνεία. Το άρθρο 90, παράγραφος 6 του κανονισμού, καθορίζει τη συγκεκριμένη διαδικασία για την απόφαση του δικαστηρίου διακόπτει ο πρόεδρος λέει δεν είναι η παράγραφος 6, είναι η παράγραφος 7. Καθορίζει λοιπόν μια συγκεκριμένη διαδικασία για την ε, διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει το Κοινοβούλιο για την ε, απόφασή του να ζητήσει βάσει του άρθρου 128 παράγραφος 11 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γνωμοδότησε για τη δυνατότητα να συναυθεί η διεθνή συμφωνία η οποία θα συνάδει και με τις συνθήκες. Υπάρχει και ο γενικός κανόνας που προβλέπεται στο άρθρο 128 και ο γενικός κανόνας λέει ότι όταν πρόκειται να προασπίσουμε τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον ενός οργάνου της δικαιοσύνης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δηλαδή, και ο κανονισμός δεν καθορίζει ρητός ε, μια συγκεκριμένη διαδικασία, η διαδικασία που προβλέπεται το άρθρο 128 εφαρμόζεται αναλογικώς. Άρα η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να ερμηνεύσουμε και να απαντήσουμε όσον αφορά τις ε, συμφωνίες που δεν αναφέρονται στο άρθρο 128, δηλαδή ε, να ισχύει το άρθρο 90. Όσον αφορά τις υπόλοιπες πράξεις οι οποίες δεν αναφέρονται στο άρθρο 128, αλλά η επανεξέτασή τους ε, για τη δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο όπως και στις υπόλοιπες πράξεις θα πρέπει να εφαρμόζεται μια ερμηνεία λογική και να θεωρήσουμε ότι συμπεριλαμβάνονται και αυτά στη γενική διαδικασία του άρθρου 128. Αν θέλει κάποιο το λόγο μπορεί κάλλιστα να αναλάβει το λόγο, αλλά προφανώς αυτά ισχύουν. Ο κύριο Νταφ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως με την ερμηνεία που δίνεται για την παρούσα κατάσταση. Συμφωνώ μαζί σας. Και μάλιστα εγώ ζήτησα από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να ζητήσουμε ε, την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αλληλευτική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου που θεωρώ ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υπάρχει ένα κενό στους ε, κανόνες που σημαίνει ότι τα επόμενα βήματα του Προέδρου είναι αβέβαια. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε τη δυνητική χρήση του άρθρου 90 σε αυτή την περίπτωση. Χρειάζεται απαρτία για να αποστείλετε εσείς επιστολή. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι και λίγο επαχθής διαδικασία. Θα, νομίζω ότι θα μπορούσατε κάλλιστα να αποστείλετε την επιστολή στον Πρόεδρο. Κύριος Χέφνερ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Καταρχάς, σας ευχαριστώ γιατί θίξατε το ζήτημα αυτό και το έχετε συμπεριλάβει στην σημερινή διμερήσια διάταξη κατόπιν ετήσιός μου και Κατά δεύτερον, σας ευχαριστώ διότι εξετάσατε εντελεχώς την πρόταση και μας παρουσιάσατε την άποψή σας. Το θέμα προκύπτει από μια διαφορά σε τροπολογία της ομάδας μου σε άλλη επιτροπή του Κοινοβουλίου. Και ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε και εδώ διότι είμαστε Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια ερμηνεία στο ζήτημα. Μπορώ να σας πω ότι για την απάντηση που μας έχετε ε, δώσει συμφωνώ απολύτως η δυνατότητα να αποστείλουμε αυτή την επιστολή. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να φροντίσουμε οι διατάξεις του κανονισμού να ερμηνεύονται όσο το δυνατόν σαφέστερα και νομίζω ότι ε, σε αυτό συμφωνούμε όλοι εδώ στην Επιτροπή μας. Ζήτησα επίσης να ε, εγγραφεί το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη, όχι γιατί είχα κάποια αμφιβολία για την ε, πιθανή ερμηνεία, αλλά για να προχωρήσει η διαδικασία. Διότι θα ήταν λίγο δυσάρεστο αν σήμερα δεν μπορούσαμε να δώσουμε στην Επιτροπή μία απάντηση η οποία να είναι και πλέον κατάλληλη. Ε, εσείς πλέον είστε αρμόδιος για να αποφασίσετε πότε, ε, πόσο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε το θέμα ώστε να δώσουμε μια απάντηση ως Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν. Ο κύριος Νταφ, ε, διαδικαστικό ζήτημα. Πόσα άτομα είναι η απαρτία για την Επιτροπή. Γνωρίζει κανείς. Το 1 τέταρτο λέει ο Πρόεδρος. Όπως γίνεται συνήθως, εγώ φταίω, διότι κατά κανόνα ο αριθμός αποτελεί πρόσκομα αν ζητήσει κάποιος να επαληθεύσουμε ότι έχουμε απαρτία. Και τελικώς εγώ ήμουν ο πρώτος ο οποίος ε, έκανε λάθος και το έθεσα μόνο μου το ζήτημα. Δεν το είχε ζητήσει και κανείς. Ε, κύριε Χέχνερ, αλλάζει τίποτα εάν ληφθεί απόφαση να αποσταλεί επιστολή την επόμενη, στην επόμενη συνεδρίαση. Πότε την επόμενη συνεδρίαση? Είναι την επόμενη εβδομάδα, στις 22 του μηνός. Έχουμε ήδη αποφασίσει ότι θα κάνουμε μια εκτακτή συνεδρίαση. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να απαντήσουμε επισήμως στις 22. Κατά την άποψή μου, προλαβαίνουμε. Δεν ξέρω αν εσείς, ε, γράφοντας αυτή την επιστολή, Ίσως θα έπρεπε να έρθετε σε επαφή και με τον συντονιστή του ΕΛΚ. Δύσκολα βέβαια θα μπορούσα να πιστέψω ότι κάποιο μέλος της Επιτροπής μας δεν θα ήταν αντίθετο. Η απαρτία απλώς μας επιβεβαιώνει ότι μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να αμφισβητεί την απαρτία. Παρά το γεγονό ότι εσεί αναφερθήκατε στην απαρτία, κανένα δεν ζήτησε να επαληθεύσουμε ότι έχουμε απαρτία. Επομένω, ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε και σήμερα να λάβουμε την απόφαση. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σα, ναι, και στι 22 να ψηφίσουμε, πάλι προλαβαίνουμε. Ωραία. Θα ψηφίσουμε στι 22. Η ανακοίνωση στην Ολομέλεια θα γίνει στι 23. Ε, κύριε Γκερέρο. Ήθελα απλώ να υποστηρίξω την πρότασή σα να λάβουμε απόφαση στι 22 του μηνό, διότι ναι μεν ε, είναι ελάχιστε μέρες, αλλά από την άλλη το να μην ρωτήσουμε αν έχει απαρτία ε, είναι ιταλική λύση, αλλά μπορεί να υπάρχει και γερμανική ερμηνεία του ζητήματος ή ισπανική ερμηνεία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές πολιτικές ομάδες που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση και δεν είναι τόσο κατεπήγον ε, το θέμα. Μπορούμε να περιμένουμε κάλλιστα μια εβδομάδα πριν αποφασίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι πιο λογικό θα ήταν να περιμένουμε λίγες μέρες και ίσως θα ήταν και χρήσιμο να Έχουμε γραπτό στην ε, πρόταση που κάνατε και προφορικός. Αλλά μόνο εδώ ενώπιόν μας σήμερα προφορικός την κάνατε. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάποιες μέρες και να ε, ψηφίσουμε την επόμενη φορά. Καλώς. Ωραία, λοιπόν. Θα το ξανασυζητήσουμε στις 22 του μηνός. Ε, θα πρέπει να ε, είμαστε σε επαφή όλοι. Εγώ μετά από πρόταση της γραμματείας που γνωρίζει πολύ καλύτερα τα πράγματα από μένα, αλλά σας το λέω και εγώ, ο κανονισμός ε, απαιτεί επαλήθευση της απαρτίας. Σε ποιο άρθρο είναι? Άρθρο 195 παράγραφος 2. Δεν είναι ούτε Ιταλική, ούτε Ισπανική, ούτε Γερμανική λύση λοιπόν. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Θα πρέπει να πω ότι ζητήθηκε έκτακτη συνεδρίαση στις 7 Απριλίου νομίζω. Ναι. Στις 22 Μαρτίου και στις 7 Απριλίου έχουμε έκτακτες συνεδριάσεις και έγινε δεκτείο. Νομίζω δεν έχουμε να αποφασίσουμε κάτι άλλο. Η προσεχή συνεδριάση είναι για τις 18 και 19 Απριλίου. Ούτως ή άλλως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι πιο πολλές οι έκτακτες συνεδριάσεις από τις ε, τακτικές. Ένδειξη ότι εργαζόμαστε όλοι. Ευχαριστώ. Είστε πανηδί.